Yes, hello. Welcome. We will start the meeting Grotis, a little bit coming later today. Καλησπέρα σας, σας ξεκινήσουμε. Ο... Εγώ θα ε, προεδρεύσω προς το παρόν, ο κύριος Γερμπράντη θα αναλάβει στις 5 ε, παρατέταρτο. Ε, προτείνω να κάνουμε δύο αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Το 18 για την ε, πρόσβαση στους γενετικούς χώρους και δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφειλών. Ε, μας ζήτησε η κυρία Μπελιέ να το αναβάλουμε και θα το συζητήσουμε στην πρώτη συνεδρίαση του Ιανουαρίου. Μετά έχουμε ένα νέο σημείο στα διάφορα. Επισήμανση του ε, κρέατος ε, από τον κανονισμό για τα τρόφιμα, αρθή 28α και 17 17 Δεκεμβρίου θα γίνει η συζήτηση αύριο στις 12 λοιπόν με εκπροσώπους της Κομισιόν. Και επίσης έχουμε όλες τις ε, γλώσσες ε, εκτός από Μαλτέζικα και Εσθονικά και άλλη μια ανακοίνωση. Ο κύριος Γιώργενσεν ορίστηκε ε, Υπουργό Γεωργίας και αλληλία στην Δανία. Μας αφήνει λοιπόν, αλλά πάει σε μια καλή και πολύ ενδιαφέρουσα θέση του ευχόμαστε καλή επιτυχία, γιατί το πρώτο θέμα που θα έχει να αναλάβει είναι οι ποσοστώσεις. Μετά, για την ε, ευζοία των ζώων και για τα ζυζανιοκτώνα, οι ψηφοφορίες πάνε για τις 22 Γενάρη. Ε, τροπολογίες για, για το πολυπλασιαστικό υλικό, αναπαραγωγικό υλικό, ε, πάει για τις 18 Δεκέμβρη στις 12 το μεσημέρι. Και βεβαίω όλα αυτά θα συζητηθούν 30 Γενάρη του χρόνου. Μετά. Τριμερής διάλογος. Θωριούχα αέρια, 16 σήμερα, από τις 2 μέχρι τις 5 ο πρωί ο διάλογος. Πρόσβαση ε, στις, στα προνοιακά επιδόματα έκθεση Μπελιέ έχει καθυστερήσει, θα πάει το Γενάρη η ψηφοφορία και η ενίσχυση των υποχρεώσεων των χρηστών. Μετά έχουμε τον, καπνό, την έκθεση Μακέβαν, θα συναντηθούμε απόψε. Έχουμε ένα τέταρτο τριμερή διάλογο, στις, είχαμε ένα τέταρτο τριμερή διάλογο στις 11 ε, Δεκέμβρη. Έχουμε προχωρήσει με το Συμβούλιο, πρέπει να πω. Οπότε ελπίζω απόψε το βράδυ να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Προσπαθούμε όλοι να καταλήξουμε σε μια συμβαστική πρόταση για τις κλινικές δοκιμές η συνολική, ευρέθη η συνολική α, συμφωνία στο Στρασβούργο στις 12 και οι τεχνικές συζητήσεις συνεχίζονται για να ολοκληρωθεί το κείμενο, το οποίο θα παρουσιαστεί στην Κορεπέρ και στην Επιτροπή. Η, α, η Λιθουανική Προεδρία θέλει να πάει στις 20 Δεκεμβρίου στην Κορεπέρ με το θέμα αυτό. Επίσης, ε, υπήρξε μια συμφωνία για τα βιοκτώνα α, στις 2 Δεκεμβρίου και για την Ευρω... Ε, περιβαλλοντική αξιολόγηση επιπτώσεων ο δεύτερος και ο τρίτος τριμερής διάλογος έγινε στις 26 Νοεμβρίου και στις 11 ε, Δεκέμβρη. Συγγνώμη. Και ο πρώτος ε, τριμερής διάλογος θα γίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Γενάρη, οπότε έχουμε αρκετούς διαλόγους, τριμερείς διαλόγους που ε, τρέχουν ακόμη, βεβαίω θα ολοκληρωθούν και κάποιοι. Έχουμε το εργαστήριο για τα χωροκατακτητικά είδη αύριο στις 12.30 με ε, τις 3.30. Ε, στο 3 g 3 Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Γκρότε, για να, αφού ήρθε, να αναλάβει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Είμαστε στο σημείο 3 και τι έκπληξη, είμαστε στην έκθεσή μου. Προστασία των ειδών άγριας πανίδας χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους. Να περάσω στα γερμανικά. Ε, τυπική αυτή η έκθεση που <laughs> μένει για τον πρόεδρο να την αναλάβει. Ε, θυμάμαι και την ε, μετάβαση στην ε, ε, Λισαβόνα που μας υποχρεώνει να κάνουμε αυτή την αδιατύπωση για να δούμε τι κάνουμε με την επιτροπολογία. Δεν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές, ούτε τροπολογίες ουσιώδεις. Έχουμε 13 ε, τροπολογίες οι οποίες έχουν ως στόχο αυτές οι εκτελεστικές ε, ε, πράξεις να αποδυναμωθούν και το, να οριστεί καλύτερα το πεδίο εφαρμογής. Αυτό είναι το πνεύμα αυτών των, αυτής της έκθεσης και των 13 τροπολογιών που έχω θέσει. Βλέπω συνάδελφος Σανώνη είναι εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, ο Σκιώτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπατε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το εμπόριο αυτών των άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας θα είναι τουλάχιστον περιορισμένο ή θα μπορεί να μειωθεί. Χρειαζόμαστε βεβαίως περισσότερες διατάξεις γιατί όλο και περισσότερα ήδη απειλούνται με εξαφάνιση και χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ελέγχους στα τελωνία. Αλλά βεβαίως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί για την απάντηση, την μόνη απάντηση στο πρόβλημα. Όπως είπατε και εσείς, η αναδιατύπωση προκύπτει ε, μετά από τον, ε, όσα λέει η κύκλη του site είναι σωστές και λόγω της Λισαβόνας πρέπει να ε, επικαιροποιήσουμε τις διατάξεις έτσι ώστε να συνάδουν με την, με την συνθήκη της Λισαβόνας κυρίως ό,τι αφορά τις κατεξοδότητες πράξεις και τις εκτελεστικές διατάξεις. Αυτό λοιπόν το θέμα είναι πολύ σημαντικό. το να δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξουσία των την, να υιοθετεί ε, κατεξοδότηση πράξης σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατική νομοποίηση για το Κοινοβούλιο. το 5, 6, 8 και 9 οι τροπολογίες δηλαδή δίνουν την, τις εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Κομισιόν και νομίζω ότι βασίζονται στην σωστή νομική βάση. τα έγγραφα που θα γίνουν, ε, που, θα, που αφορούν τις κοινοποιήσεις δηλαδή και τα πιστοποιητικά Ως ε, σκιώδης λοιπόν από την ομάδα μου, εγώ πραγματικά θα προτείνω την υποψήφιση της έκθεσης στην ομάδα. Ευχαριστώ. Πολύ χαίρομαι, αυτό θέλουμε κι εμείς από τους φιλελεύθερους, να μας υποστηρίξουν. Πάμε παρακάτω. Η κυρία Χάση δεν είναι εδώ. Δεν έχουμε άλλες παρεμβάσεις. Η Κομισιόν είναι παρούσα. Παρακαλώ, να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν ή την εκπρόσωπο. Thank you, Mr. Chair. Uh, I think... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και εσείς εξηγήσατε, το έγγραφο αυτό αποτελεί αναδιατύπωση κανονισμού που υιοθετήθηκε εδώ και αρκετό καιρό και που έχει τροποποιηθεί επανειλημμένος, κυρίως στα παραρτήματά του, ε, για να προσαρμοστεί στην διάσκεψη των ε, συμβαλωμένων της ε, Σύμβασης ΣΥΤΕΣ η Κομισιόν ε, πρότεινε να ευθυγραμμιστεί και με τις διατάξεις επιτροπολογίας που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας υπό το πνεύμα ε, της προηγούμενης διαδικασίας επιτροπολογίας ε, προσαρμοσμένης βέβαια στις καινούριες διατάξεις της συνθήκης Λισαβόνας. Λάβουμε υπόψη την έκθεση, το σχέδιο έκθεσης ε, και ελπίζω ότι στο Συμβούλιο θα επιτευχθεί συμφωνία τι επόμενε εβδομάδε ή μηνες για αυτό το έγγραφο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ωραία. Η ε, παθισμια για τις τροπολογίε τροπολογίες είναι η 7η Ιανουαρίου ε, και στην, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 30 Ιανουαρίου. Πάμε στον Ραβόσιτο σύμφωνα με την οδηγία 2018 έχουμε εδώ μια παρέμβαση από την κυρία Χάση, από την Dagmar Ροντμπέρεν, τον κύριο Σανώνη, δεν ξέρω τώρα ποιος ακριβώς θα πάρει το λόγο, ο κύριος Στάς. Ε, ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. δέκα μέλη από όλες τις πολιτικές ομάδες διαφωνούν στεναρά με την πρόταση της Κομισιόν για αυτό το τύπο αραβόστου, αυτό το στέλεχος. Ελπίζουμε ότι ε, θα πείσουμε με τα πολύ λεπτομερή μας επιχειρήματα για το ε, πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, έχει προσαρμόσει την οδηγία 2018. Ε, πιστεύουμε ότι δεν τηρούνται, παραβιάζονται διάφορα άρθρα αυτής της βασικής οδηγίας. Και δεν συμφωνούμε επίσης και με τον ορισμό κάποιων γεωγραφικών ζωνών η Επιτροπή Ασφάλειας των Τροφίμων δεν εξέφρασε γνωμοδότηση, αλλά έγινε συζήτηση εκεί για το θέμα αυτό και από τότε που έγινε η πρώτη πληροφορία, η Επιτροπή αυτή εξέδωσε τρεις γνωμοδοτήσεις για το σύνολο του θέματος ε, σε, ε, επί τη βάση αυτών των ε, ε, των γνωμοδοτήσεων και από τη βάση της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλισης των Τροφίμων η Κομισιόν άλλαξε την πρότασή της, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ακόμα και η τροποποιημένη πρόταση ε, δεν ε, ακολούθησε τη σωστή διαδικασία. Πριν υποβληθεί στους Υπουργούς έπρεπε να έχει υποβληθεί στην Συμβουλευτική Επιτροπή η Κομισιόν έχει υπερβεί τις αρμοδιότητές της και τις εξουσίες που της έχουν παραχωρηθεί. Έχουμε και, είχαμε και στο παρελθόν ένα παρόμοιο ζήτημα με την, ε, την πρόταση της Κομισιόν για την κυκλοφορία ενός συγκεκριμένου είδους πατάτας η οποία ακυρώθηκε από το ε, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το εκτιμώντας ρο, ε, έκανε αναφορά στην ε, άδεια που θα είχε, μπορούσε να έχει δώσει η Κομισιόν για αυτό το είδος πατάτας. Ε, ε εμείς αυτό το σε αυτήν την παράγραφο ε, αναφερόμαστε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της περασμένης εβδομάδας. Η ε, Υπηρεσία Ασφάλισης των Τροφίμων ε, πρέπει να κάνει μια πλήρη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάνουμε αναφορά και στην συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση της έκθεσης Λεπάζ η οποία όμως δεν έχει προχωρήσει στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ. Η κατάσταση στην ε, Επιτροπή για τους γενετικά στροποποιημένους οργανισμούς δεν αντικατοπτρίζει την κατάσταση στον, ε, στην πλειοψηφία των κρατών μελών. Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Και νομίζω ότι δεν αδικό κανένα. Ούτε τον Ερικ Πουντελέ ούτε τους συναδέλφους, ούτε κανέναν από τις διάφορες γενικές διευθύνσεις. Όταν λέω ότι στην Κομισιόν η ευαισθησία για την απελευθέρωση ενό τέτοιου γενετικό ορπημένου οργανισμού δεν είναι ιδιαίτερως αυξημένη. Αυτό μάλλον έχει να κάνει με το ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Κομισιόν και το ανώτατα κλιμάκια έχουν άλλα διαφορετικά, ίσως πιο σημαντικά θέματα να ασχοληθούν και αυτό το σέβομαι. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει τελικά μια απελευθέρωση ενό τέτοιου οργανισμού. Δέχομαι ότι τις προηγούμενες εβδομάδες ε, μετά την απόφαση του ε, δικαστηρίου ε, αποσύρθηκα λίγο και είπα ναι, τελικά δεν είπε τίποτα το δικαστήριο. Ήταν επί της ουσίας λάθος η απόφαση για τις πατάτες, αλλά η Κομισιόν, είπε το κοινοβούλιο, είπε μάλλον το δικαστήριο συγγνώμη, ότι η Κομισιόν έκανε λάθος. Και μίλησα με τον κύριο Νταλή και μίλησα και του είπα τι ακριβώς, τι ακριβώς κάνετε. Λάθος είναι αυτή η απόφαση. Υπάρχει ένας λόγος. Ότι δεν υπάρχει ευαισθησία. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα νομικά της υπόθεσης. Το δικαστήριο ε, ζήτησε από την ε, Κομισιόν σε περίπτωση που ε, υπάρχει αυτό το εκρεμές παράρτημα για το να τον το να κάνει κάτι. Το δικαστήριο δεν είπε ότι πρέπει να το επιτρέψει. Είπε ότι η Κομισιόν κάτι πρέπει να κάνει το Σεπτέμβριο. Οπότε η Κομισιόν θα μπορούσε να αρνηθεί την απελευθέρωση. Τώρα σήμερα ακούμε ποια είναι η πρόταση της Κομισιόν. Ε, εμένα το, κανονικά θα έπρεπε να πούμε όχι. Αυτό μου λέει το ένστικτό μου για αυτό το... Ε, τον Αραβό στο 1507. Έχουμε και τη γνωμοδότηση της ε, ΕΦΣΑ. που είναι αρκετά ε, αρνητική, όπως και για την Ασπαρτάμι, θα τη δούμε αύριο. Και έχουμε και μια δημόσια συζήτηση για την απελευθέρωση γενικώ, συνολικώς. Και έχουμε και επιστημονικές ε, ε, μελέτες, στοιχεία, μας που λένε ότι αυτός ο αραβός του 1507 είναι, αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία. Βεβαίως θα ακουστούν όλα τα επιμέρους επιχειρήματα. Βεβαίως ε, αυτό το... Ε, ε, αυτό το, αυτός ο ραβόστος έχει λέει ότι επειδή ακριβώς είναι γενετικός τροποποιημένος είναι, μπορεί να καταστρέψει κάποιες επιζωτίες, να τις ακυρώσει. Εντάξει, έχουμε, έχει δίκιο ο συνάδελφος, θα πρέπει η, ε, έκθεση να αντικατοπτρίζει τα όσα λέει και η απόφαση του ε, δικαστηρίου, αλλά πρέπει η Κομισιόν να τα λάβει υπόψη της αυτά. Έξι κράτη-μέλη είναι ιδιαίτερως ε, συντηρητικά απέναντι σε αυτή την απόφαση. Και επίση ξέρουμε το μεταξύ ότι δεν υπάρχουν νέε αιτήσει για απελευθέρωση. Πρέπει η Κομισιόν να ψάξει για να βρει. Νομίζω λοιπόν ότι το ψήφισμα που έχουμε υποβάλει είναι καλό. και δίνει νομίζω το σωστό μήνυμα για το τι πρέπει να φτάσει προς τα έξω, προς τους πολίτες μας, αλλά και τα, και τα κυρία Λεπάζου. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τους συναδέλφους. Συμφωνώ απολύτως και με αυτά που είπαν η κυρία Ροκπέρεντ και ο κύριος Στάς. Υπάρχουν πάρα, πολλές, πάρα πολλοί λόγοι ε, Υπερψήφιση του ψηφισματό μα και απόρριψη αυτού του αιτήματος. Ε, τακτός ή άλλως εμείς ε, σύμφωνη γνώμη μπορούμε να δώσουμε. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να εκφράσουμε την διαφωνία μας, το οποίο σε, πολιτική, σε πολιτικό επίπεδο είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο μπορούμε λοιπόν να λάβουμε αυτή τη θέση, το είπατε. Οι μελέτες είναι ότι υπάρχουν, είπαν ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στα ε, λεπιδόπτερα, παρά το γεγονός ότι η ΕΦΣΑ δεν έκανε τις συμπληρωματικές μελέτες που χρειάζονταν για να δείξει ακριβώς τι χρειάζεται για να, επιλύσουν, για να επιληθούν τα προβλήματα που τίθενται. Ζητήσαμε ενίσχυση της αξιολόγησης ε, των γενετικώς ε, τροποποιημένων οργανισμών. Δεν έχουμε τις σχετικές μελέτες. Πριν από δύο χρόνια ψηφίσαμε βάσει πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με μεγάλη πλειοψηφία βέβαια κόλλησε ο φάκελος εδώ και δυόμιση χρόνια στο Συμβούλιο και το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ε, να δοθεί αυτή η έγκριση. Όσον αφορά το επιχείρημα ότι το δικαστήριο θα είχε επιβάλει κυρώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δεν είχε δώσει την ε, έγκριση. Όχι. Το γεγονός ε, που είναι άξιον κύρωσης είναι το γεγονός ότι δεν τοποθετηθήκαμε η εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης ε, μπορεί να ε, σημαίνει απόρριψη, δεν σημαίνει υποχρεωτικά έγκριση και νομίζω ότι είναι πολύ πιο δικαιολογημένη μια τέτοια απόρριψη. Συμφωνώ απολύτως ότι ε, το σκεπτικό του δικαστηρίου σε σχέση με την ποικιλία πατάτας φλόρα το εξηγήσαμε πάρα πολλές φορές, το είπαμε πολλές φορές, αν φλόρα, ε, είπαμε πάρα πολλές φορές λοιπόν ότι η έγκριση ήταν παράνομη γιατί δεν είχε ε, υπάρξει διαβούλευση με όλα τα κράτη-μέλη εκ νέων. Κατά τη γνώμη μου, ε, αν υπήρξαν νέε μελέτε, δεν υπήρξε διαβούλευση νέα με τα κράτη-μέλη. Επομένω, όλα συγκλίνουν προ την πρόταση, που, τη θέση που θέλουμε να λάβουμε δηλαδή απόρριψη αυτής της έγκρισης ε, στο πλαίσιο της επιτροπολογίας. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάνκη. Αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνώ 100% με την άποψη που εξέφρασαν οι συνάδελφοι. Πρέπει να έχουμε μια σωστή, συγκεκριμένη απόφαση για αυτούς τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τις συνέπειες που έχουν στην ανθρώπινη υγεία. Ε, ο τομέας αυτός έχει τύχει ιδιαίτερα μεγάλη έρευνα στα τελευταία χρόνια και πρέπει και εμείς να λάβουμε μια θέση ή να ξανασκεφτούμε τη θέση μας απέναντι σε αυτά τα φυτά. Είναι συγκεκριμένη λοιπόν η άποψή μας, γιατί ε, η Ουγγαρία, και το λέει το Σύνταγμά μας, αποκλείει και απαγορεύει την ε, καλλιέργεια τέτοιων γενετικώς τροποποιημένων φυτών. Οπότε και εμείς ε, ε, ανησυχούμε και ελπίζουμε ότι και οι γειτονικέ μας χώρες θα λάβουν τέτοιες αποφάσεις. Βεβαίως και το Κοινοβούλιο πρέπει να στείλει ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Δεν πρέπει να δοθεί πράσινο φως στην Κομισιόν. η Κομισιόν έχει κάνει λάθος με αυτή την υπόθεση, κυρίως όταν ενέκρινε τις πατάτες. Και αν, ε, προχωρήσουμε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε συγκεκριμένα και προσεκτικά και συντηρητικά, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα είναι πλεονέκτημα για μας αυτά τα φυτά να μην τα προωθήσουμε στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Μπάνκι. Thank you. Well, usually Ευχαριστώ κυρία Γκέρλινγκ. Μου συμβαίνει συχνά σε τέτοιου από συζητήσεις να έχω την αντίθετη άποψη. Εγώ πιστεύω ότι όλες μας οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε στοιχεία ε, σε επιστημονικά στοιχεία όπως μας παρουσιάζονται και όπως ε, μας ε, διοχετεύονται από τις υπηρεσίες που τις πληρώνουμε πολύ ακριβά για να κάνουν αξιολογήσεις εκ μέρους μας και όχι για λόγους ιδεολογικούς συλλήβδιν να απορρίπτουμε τέτοιου είδους άδειε και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε γενικές ε, γραμμές ε, η έγκριση γενετικώς τροποποιημένων ε, οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντικείμενο μιας πολύ αυστηρής διαδικασίας και λέμε ότι εντάξει καλό θα ήταν ίσως να απορρίψουμε την άδεια αυτή βέβαια το θέμα του αραβοσίτου της Μονσάντο δεν είναι κάτι το οποίο μεμονωμένα αντιμετωπίζεται γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ε, ε τις διαδικασίες, ε, τι σχέση έχει η πατάτα με τον αραβόσιτο εμπροκειμένο. Αυτό που έχουμε εμπροκειμένο μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε είναι μία άδεια ενός προϊόντος ή όχι. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε πολύ ε, σοβαρούς και συγκεκριμένους επιστημονικούς λόγους να απορρίψουμε την έγκριση αυτή. Εγώ δεν άκουσα κανέναν σοβαρό επιστημονικό λόγο και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι λόγοι κατά τη γνώμη μου. Νομίζω ότι είναι γεγονός ότι το δικαστήριο κατέκρινε την ε, καθυστέρηση των αποφάσεων, όχι τις ίδιες αποφάσεις και ο λόγος καθυστέρησης απόφασης είναι ότι το πρόβλημα είναι μια αδιάλακτη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για το θέμα αυτό. Η ΕΦΣΑ έχει επιμείνει στα επιστημονικά στοιχεία και δεν μπορεί να υποστηρίξει την άποψη του Κοινοβουλίου επί της βάσης αυτής δεν πηγαίνουμε πουθενά, κάτι το οποίο βέβαια βολεύει τους περισσότερους ε, σε αυτή την αίθουσα. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ, γιατί ουσιαστικά δεν νομίζω ότι δημιουργούμε κανένα συγκριτικό πλεονέκτημα για μας, το αντίθετο κάνουμε και οι προκλήσεις ε, για τη γεωργία, για την ε, παραγωγή, για την αποτελεσματικότητα είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορούμε να ε, αγνοήσουμε μια τεράστια, μια ολόκληρη τεχνολογία κατά αυτόν τον τρόπο. Προφανώς είναι, είναι η μειοψηφία στη συγκεκριμένη επιτροπή, αλλά θα ήθελα να ακουστεί και η δική μου άποψη θα καταβάλω όση προσπάθεια περνάει από το χέρι μου για να μην καταψηφιστεί η ε, έγκριση αυτή. Δεν είναι δυνατόν ε, να λέτε ότι ακούτε τα επιστημονικά στοιχεία και τα λαμβάνετε υπόψη όποτε σας βολεύει και επιλεκτικά πρέπει να το κάνουμε με συνέπεια. Δεν έχουμε ξανακούσει τέτοια ομιλία για την ΕΦΣΑ. Λοιπόν, η Κομισιόν έχει τώρα το λόγο. Είναι η σειρά της. Oui, merci, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν να σας μιλήσω για την πατάτα αμφλόρα. Αληθεύει ότι η απόφαση του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη Παρασκευή ε, μας οκάρισε, μας ε, ξέπληξε. Δεν το, την αναμέναμε. Όμως ε, αναλύοντας το σκεπτικό αυτής της απόφασης είναι σημαντικό να μπορέσουμε να κάνουμε τη διάκριση με τον Αραβό στο 1507. Για την πατάτα το δικαστήριο μας καταδίκασε διότι αφού υποβάλαμε την απόφαση για την αμφλόρα στο Συμβούλιο η Κομισιόν δεν υιοθέτησε αμέσως την απόφαση για την αδειοδότηση της καλλιέργειας της αμφλόρας. Το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η ΕΦΣΑ υπέβαλε μια νέα επιστημονική γνωμοδότηση με δύο μειοψηφούσες γνώμες, α, ψήφους, την οποία πήραμε υπόψη, διότι ε, την απηχήσαμε σε ε, παραγράφους αιτιολογικής έκθεσης, αλλά το δικαστήριο είπε ότι θα έπρεπε να έχουμε επιστρέψει στη μόνιμη επιτροπή και, να, και να, θα έπρεπε να έχουμε ξαναξεκινήσει τη διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο μας καταδίκασε το δικαστήριο. Εδώ για τον Αραβό το 1507 η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Σας υπενθυμίζω ότι το πρώτο αίτημα κατατέθηκε το 2001. Έκτοτε ε, η ΕΦΣΑ έξι φορές νομοδότησε θετικά. Η Κομισιόν για ε, δύο φορές παραλίγο να καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για καθυστερήσεις. Τελευταία φορά το 2013. Για αμέλεια μάλλον, όχι για καθυστερήσεις. Για αμέλεια να θέσουμε το κείμενο υπόψη του Συμβουλίου. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας καταδίκασε διότι παρόλη την ψηφοφορία της ε, Μόνιμης Επιτροπής το 2009 που δεν έλαβε δική πλειοψηφία, η Κομισιόν ε, δεν απέστειλε το σχέδιο αυτό στο Συμβούλιο από το 2009 και μετά όπως προβλέπουν οι διαδικασίες. Δεν θα μας ικανοποιούσε να στείλουμε το κείμενο της Αμόνιμης Επιτροπής του 2009 στο Συμβουλίο, γιατί η ΕΦΣΑ το 2000, ε, μέχρι το 2012, μάλλον το 2012, εξέδωσε δύο καινούς νομοδοτήσεις για το 1507, δύο καινούς νομοδοτήσεις οι οποίες καθησύχαζαν ε, τις προηγούμενες ανησυχίες και ε, τις προηγούμενες τέσσερις εκθέσεις της ΕΦΣΑ. Είναι αλήθεια ότι Είχαμε ζητήσει από την εταιρεία να ξαναυποβάλει το φάκελο για να λάβει υπόψη την ομοδή της ΕΦΣΑ. Η Pioneer, η εταιρεία αυτή, δεν μας ικανοποίησε αυτό μας το αίτημα. Όμως, κατόπιν της απόφασης του δικαστηρίου, το Σεπτέμβριο 2013, η Pioneer μας επιβεβαίωσε ότι θα προσάρμοζε ε, το ε, σχέδιο παρακολούθησης έτσι ώστε να το εφηγραμμίσει με τις τελευταίες συστάσεις της ΕΦΣΑ. Συνεπώς, όπως και το προβλέπει και η πρόταση που υποβάλαμε στο Συμβούλιο, το πρόγραμμα αυτό, το σχέδιο αυτό θα συζητηθεί με τα κράτη-μέλη. Ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν έφυγε σήμερα αλλά είχε φύγει παλιότερα, η πραγματική αντίσταση στο ε, γλουφοσυνικό αμμόνιο που ε, είναι παραστοκτόνο, αλλά είχε συμπληρωθεί στο αρχικό αίτημα της Pioneer. Ε, το παραστοκτόνο όμως αυτό δεν έχει αδειοδοτηθεί για τον, καλα... για τον συνεπώς δεν θα χρησιμοποιηθεί. Αν ο αραβόστος αυτός λάβει άδεια ε, καλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το γλυφοσυνικό αμμόνιο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον αραβόστο. Αν ένας γεωργός αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το απόθεμα γλυφοσυνικού αμμονίου που του έχει χορηγηθεί για, άλλους, για άλλες καλλιέργειες, αυτό θα ήταν αδίκημα και θα μπορούσε να τιμωρηθεί. Ε, η πρόταση ψηφίσματό σα αναφέρεται στην ανάγκη επίσης να λάβουμε υπόψη τα μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα συνέπειες ε, των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και σε οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι στόχο τους, όπως για παράδειγμα αυτά τα περίφημα λεπιδόπτερα. Γι' αυτό το λόγο στην πρόταση απόφαση που αποστήλαμε στο Συμβούλιο έχουμε προσθέσει ε, μέτρα για να περιορίσουμε στο μέτρο του ε, δυνατού την επίδραση σε τέτοιου είδου ε, οργανισμούς. <clears throat> Θεωρούμε ότι εφαρμόσαμε πλήρως την αρχή της πρόληψης ε, σε ό,τι αφορά την προστασία των εντόμων τα οποία δεν είναι στόχος του, ε, του αραβόστου αυτού. Επίσης λάβαμε υπόψη το θέμα της γύρης ε, και του επικονιασμού. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα για ορισμένε νομικές πτυχές. Στο σχέδιο ψηφίσματος αναφέρεται ότι η Κομισιόν έχει υπερβεί τις αρμοδιότητες που της χορηγεί η βασική πράξη η Κομισιόν στις 8 Νοεμβρίου υπέβαλε στο Συμβούλιο αυτή την πρόταση σχετικά με την αδειοδότηση του Αραβοσίου του 1507 γιατί, επαναλαμβάνω, γιατί το δικαστήριο μας το υπέβαλε, μας υποχρέωσε να διορθώσουμε αυτή την αμέλεια. Άλλωστε και η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημιώσεις για αυτή την καθυστέρηση διότι έχασε δύο-τρία χρόνια καλλιέργειας κατόπιν τη ε, της νομοδότησης της επιτροπή Επιτροπής του 2009. Ακολουθήσαμε σχολαστικά, με κατόπιν ε, νομικής αλλά και πολιτικής ανάλυσης, την απόφαση του δικαστηρίου. Μην ξεχνάτε ότι ε, το, η Ολομέλεια των Επιτρόπων, το κολέγιο, αποφάσισε να προωθηθεί αυτή η πρόταση προς το Συμβούλιο. Συνεπώς δεν πιστεύουμε ότι υπερβαίνουμε τις αρμοδιότητές μας. Τα κράτη-μέλη διαθέτουν τρεις μήνες προκειμένου να λάβουν απόφαση, όπως γνωρίζετε. Η ελληνική προεδρία δεν αποφάσισε να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη διαφόρων συμβουλίων. Του Συμβουλίου, για παράδειγμα, ε, της ε, ε, περιβάλλοντος στις 13 Δεκεμβρίου και σήμερα το Υπουργείο Γεωργίας η Ελληνική Προεδρία δεν αποφάσισε να εγγράψει αυτά τα θέματα, ε, αυτό το θέμα στα, στην μέση ένταση κάποιων από αυτών των συμβουλίων ε, και η Λιθουανική Προεδρία το σκέφτεται συνεπώς ενδεχομένως ε, ε το Συμβούλιο δεν θα έχει ε, πάρει απόφαση μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου στο τέλος των τριών μηνών από νομική πλευρά λοιπόν και ξεχνώντα το δική σα που είναι πολιτική σε, σε νομικό επίπεδο, αν το Συμβούλιο δεν εκφέρει γνωμοδότηση με ειδική πλειοψηφία κατά τη πρόταση, τότε η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει άδεια καλλιέργεια ε, για τον στο 1507. Αυτέ είναι οι πληροφορίε τι οποίε είχα να σα αναφέρω, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει σε καλύτερη χρονική στιγμή την ε, συνεδρίαση αυτή, ούτε να το είχαμε παραγγείλει. Νομίζω ότι επιλέξαμε τη σωστή χρονική στιγμή για να δούμε το θέμα αυτό. Άλλος κανείς θέλει το λόγο, συνάδελφοι. Όχι. Οπότε αύριο, εδώ, στην Επιτροπή μας, θα ψηφίσουμε και αν πάει στην Ολομέλεια, θα πάει στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Στην ε, η ψηφοφορία. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και την Κομισιόν για, τα, ε, ε, για τις πληροφορίες της και πάμε στη Γιούτα Χάουγκ να μιλήσουμε για τις απαλλαγές 2012. Μόνιμη εισηγήτρια η η κυρία Χάουγκ για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πάντα τα ίδια, σχεδόν τέλο πάντων πάντα τα ίδια λέω για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ε, δημόσια υγεία, τρόφιμα, ασφάλεια τροφίμων, περιβάλλον και μέτρα για την προστασία των, για το κλίμα. Όλα αυτά τα βλέπουμε μαζί με όλες τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς που εμπίπτουν στις δικές μας αρμοδιότητες. Μιλάμε δηλαδή για 0,8% του συνολικού προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να το θυμίσω αυτό. Επίσης, να ξεθυμίσω, βλέπω ότι ενδιαφέρονται πάρα πολλοί συνάδελφοι, ενδιαφερόμαστε Γιούτα, ενδιαφερόμαστε. Ε, δεν ξέρω εκεί πίσω, στο πίσω να τι γίνεται, αλλά βλέπω ότι εκεί από την πλευρά του ελεκτικού συνεδρίου δεν υπάρχει κανένας εκπρόσωπος εδώ και την, προηγούμενο, και την προηγούμενη χρονιά το ίδιο έγινε και φέτος το ίδιο γίνεται. Ελπίζω η Κομισιόν πια να λάβει ε, θέση ως προς αυτό. Το ε, ελεκτικό συνέδριο μας, βάλει, μας βάζει όλους σε μια βάρκα, σε έναν τομέα, ε, ανάπτυξη ας πούμε της υπαίθρου, ε, αλληλεία, περιβάλλον και υγεία. Όλα μαζί σε ένα καλάθι. Αυτό λοιπόν όλο το πακέτο, αυτός ο τομέας πολιτικής, ε, μιλάει για ένα 7,9, ε, μιλάμε ότι έχει ένα 7,9% ε, ποσοστό λάθους. Σε κάθε έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου αυτό αναφέρεται. Τι γίνεται. Ε, υγεία, περιβάλλον. Αν τα δούμε συνολικά θα δείτε ότι τα, α, τα λάθη γίνονται κυρίως στην ε, ανάπτυξη πέθρου και στην ελεία, όχι στο περιβάλλον και όχι στη δημόσια υγεία. Οπότε αυτό είναι πραγματικά παραπλανητικό. Το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι έχει την απόλυτη αρμοδιότητα, την απόλυτη ουδετερότητα και ότι είναι αυτό που πρέπει να δώσει το, το Ευαγγέλιο το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι οι υπόλοιποι. 7,9% ποσοστό λάθος είναι για την ανάπτυξη πέθρου και για την πολιτική αλληλείας. Και αν δούμε και τα ποσά για τα οποία μιλούμε συνολικά, αλληλεία συν ανάπτυξη πέθρου 13,75 δις ευρώ το 2012, το έτος δηλαδή για το οποίο μιλούμε. 13,75 δις ευρώ. Εμείς με, την ε, δική μας, με το δικό μας το πρόγραμμα, το Life και την Υγεία, έχουμε... Ε, αρχίζω να τα μπλέκω. 427 ε, εκατομμύρια χρησιμοποίησε. Ε, πραγματικά είναι παράλογο αυτό που γίνεται και συνέχεια το ίδιο πράγμα συζητάμε. Και συνέχεια ε, ε, φουσκώνουν κάποια τέτοια θέματα. Δεν φταίμε εμείς για τα ποσά αυτά, ούτε για το, για το ποσοστό λάθους. Ούτε η Επιτροπή μας. για την, ε, από τη Γενική Διεύθυνση ε, ε, για το κλίμα, για το περιβάλλον και για την δημόσια υγεία τα πράγματα πάνε καλά. Δεν θέλω να ξαναπώ, να ξαναπώ σε λεπτομέρειες και να πω πάλι τα ίδια, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι τα πράγματα πάνε καλά και σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς λειτουργούν καλά. Υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να υπάρξουν μια προειδοποίηση και αναφέρονται και σε εκθέσει μου, γιατί κάτι έπρεπε να γράφουν εκεί οι εκθέσει μου. Είναι ούτω ή άλλω πολύ λίγες οι παράγραφοι για την μία ή την άλλη υπηρεσία, για τον ένα ή τον άλλο οργανισμό. Βεβαίως το ελεκτικό συνέδριο για όλους τους οργανισμούς ζητά να δοθεί η τον αλλο οργανισμο Βεβαίω το ελεκτικο Αυτό πρέπει να το πω και δικαίως ε, το πράττει το ελεκτικό συνέδριο. Ε, μερικές φορές βλέπουμε και κάποια ε, αστεία πράγματα για κάποιους οργανισμούς. Ε, ξαφνικά από κάποιον οργανισμό λείπουν laptop λέει. οποία, για τα οποία μιλούμε δηλαδή για 5.000 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό, το τραγικό. Μακάρι το πρόβλημα σε όλους τους οργανισμούς να ήταν 5.000 ευρώ. Θα ήμασταν πραγματικά όλοι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και θα μπορούσαμε να περάσουμε πολύ ωραίες διακοπές. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα στους ηγητές, τους σκιώδης. Ο κύριος Φερνάντες από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να συγχαρώ την Γιούτα Χάουγκ. Μία ακόμα φορά, είναι εξαίρετη εργασία που κάνει. Συμφωνώ κατά βάση με όλα όσα αναφέρει στην έκθεσή της. Θα έπρεπε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να προτείνουμε πράγματα για τον καλύτερο ορισμό ή επανορισμό του ρόλου των διαφόρων οργανισμών και αρχών. Γιατί, γιατί ο προπολογισμό του μειώνεται όλο και περισσότερο. Θα πρέπει να ξέρουμε τι περιμένουμε από αυτές, έτσι ώστε μετά να αποφασίσουμε ποια είναι τα επαρκή μέσα που χρειάζονται για να τα βγάλουν πέρα. Επίσης, είναι σημαντικό κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες να ε, για κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες να έχουμε το ποσοστό εκτέλεσης, απορρόφησης του προπολογισμού σε κάθε τήσια έκθεση. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι ποσοστό από τον προπολογισμό της χρησιμοποιεί κάθε υπηρεσία κάθε χρόνο. Η εκτέλεση δηλαδή του προπολογισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα πρέπει να αναφέρεται στις αιτήσεις εκθέσεις. Γιατί μας δίνει μια σαφή εικόνα του έργου που έχει επιτελεστεί. Μερικές υπηρεσίε βρίσκονται κοντά στο 100% και αυτό αποδεικνύει ότι τα, ο προπολογισμό τους είναι πράγματι στενός για την ε, ε, υλοποίηση των αρμοδιοτήτων τους. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Άννα Ρόσπαρ. Det er η θέση του ECR είναι ότι κάθε ευρώ που ε, καταναλώνουμε είναι ευρώ από τις τσέπες των φορολογουμένων. Συνεπώς οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να δίνουν λογαριασμό και θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες. Σε ό,τι αφορά τις πέντε υπηρεσίες στις οποίες, οι οποίες εμπιτούν στην αρμοδιότητά μας, ε, πιστεύουμε ότι η προτάσει απαλλαγή θα πρέπει να βασίζονται στι ε, κατευθύνσεις γραμμέ του ΩΣΑ. Θα πρέπει να ακολουθούν τα διεθνώ αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα δηλαδή. Αν κάποια υπηρεσία δεν τηρεί του κανόνε, δεν θα πρέπει να λαμβάνει απαλλαγή. Δυστυχώ όμω, εμεί εδώ εξακολουθούμε να χορηγούμε απαλλαγέ, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν είναι εντάξει θέση του ECR είναι να μην χορηγούμε απαλλαγέ σε τμήματα του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής όσο οι ε, λογιστές δεν μπορούν να υπογράψουν τις λογιστικές καταστάσεις στο σύνολό τους. Έχουμε διάφορους οργανισμούς, μεταξύ αυτών και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, οι οποίοι παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα κάθε χρόνο. Συνεπώς ε, έχει λογική να ζητάμε βελτιώσεις. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τον κατάλογο των ομιλητών. Να δώσουμε το λόγο στην Κομισιά. Υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Χάουκ για την έκθεσή της ε, όσον αφορά το γενικό προϋπολογισμό και ειδικότερα το κομμάτι του περιβάλλοντος. Ε, ως προς το ελεγκτικό συνέδριο, δεν θέλω να υπερασπιστώ το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά τα κεφάλαια της έκθεσής, της, ε, του είναι σε αντιπαραβολή με το, τα κεφάλαια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και κάθε φορά μας κάνει εντύπωση να διαβάζουμε στον τύπο ότι το περιβάλλον και η γεωργία παρουσιάζουν ποσοστό σφάλματος πολύ μεγάλο και όταν βλέπουμε τις λίγες λεπτομέρειες που μας δίνει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου βλέπουμε ότι το ποσοστό σφάλματος μεταξύ περιβάλλοντος και γεωργίας δεν είναι το ίδιο. Όπως είπε και η κυρία Χάουκ, είναι καλά τα πράγματα για το περιβάλλον, λίγο λιγότερο για ε, τα θέματα του κλίματος, που είναι μια πιο πρόσφατη δραστηριότητα ε, βέβαια, με όλους τους ε, τομείς ε, ανταλλαγής δικαιωμάτων ε, εκπομπών αερίων που αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες έβρεσης αναδόχων, εμπειρογνωμόνων σε αυτόν τον τομέα που να γνωρίζουν καλά τον τομέα και να μπορούν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία τους ζητάει η Γενική Διεύθυνση Κλίματος. Αυτά έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Γιούτα, για να κλείσουμε. Ευχαριστώ αυτό που είπε ο Χωσέ Μανουέλ, ότι πρέπει να δούμε ποιο είναι το ποσοστό του προπολογισμού ε, που χρησιμοποιείται για τη δαπάνη στον οργανισμό, μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το συμπεριλάβουμε. Ε, δεν είναι τίποτα, ένα, μια, δύο πράξεις πρέπει να γίνουν υπολογισμού. Ε, αυτό που είπε τώρα η κυρία Ρόσπαχ είναι μάλλον πιο δύσκολο να γίνει. Γιατί εγώ δεν μπορώ, εγώ ως κοινοβούλιο μιλώ τώρα, δεν μπορώ να υποχρεώσω τις, ε, τους οργανισμούς να, υπολογίζουν, ε, να κάνουν τους υπολογισμούς τους ανάλογα με τον ΩΣΑ. Ε, έχουν με βάση το βασικό κανονισμό, τον οποίο εμείς μαζί με το Συμβούλιο έχουμε, τους έχουμε δώσει, την υποχρέωση να φροντίζουν για τα δημοσιονομικά τους δυνάμει αυτού του κανονισμού. Οπότε αυτοί πρέπει να... Εμείς τους καθοδηγούμε, ο δικός μας ο κανονισμός. Τώρα για την διαφάνεια... Βεβαίως πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια και για την εργασία της κάθε, του κάθε οργανισμού, αλλά και διαφάνεια για, τον, για τις διάφορες επιστημονικές επιτροπές των οργανισμών. Νομίζω ότι εκεί όλες οι, ε, όλοι οι οργανισμοί έχουν κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο και όλα τα στοιχεία, ε, όλα τα θέματα τα οποία διαχειρίζονται οι οργανισμοί, εκεί δηλαδή που μπορούν να ορίσουν ποιο θα μπει στην κάθε επιστημονική ομάδα, ε, αυτό μπορούν να μας το έχουν δηλώσει. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε, τα έχουν πάει καλά. Αυτό για το οποίο ε, μπορούμε να παραπονηθούμε είναι η δράση της Κομισιόν για κάποια σημεία, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλο θέμα. Ας το αφήσουμε πέραν, εκτός αυτής της συζήτησης για την απαλλαγή. Σημαντική η παρατήρησή σου. Πάντα με αυτούς τους, ε, τους οργανισμούς ε, υπάρχουν διάφορες α, δυσκολίες. Βεβαίως οι οργανισμοί είναι και ανεξάρτητοι πέραν από τον άλλον. Λοιπόν, ε, προθεσμία για τροπολογίες 18 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί. 31 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε για την απαλλαγή και μετά στην Επιτροπή Προπολογισμού, Ελέγχου του Προπολογισμού, 18 Φλεβάρι θα γίνει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει 17-18 Μαρτίου στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Οπότε, κλείνουμε τα σημεία 5 έως 10 της σημερινής διάταξης και πάμε στην έκθεση του κυρίου Ποκ. Σημείο 11 λοιπόν. Yes. Ε, ευχαριστώ Ορισμένα ξένα είδη όταν ε, μεταφέρονται εκτός του περιβάλλοντος τους ε, μπορούν να αρχίσουν να εξαπλώνονται ε, χωροκατακτητικά και δημιουργώντας σημαντικές επιπτώσεις περιβαλλοντικές και οικονομικές. Οι 12 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ είναι οι ζημιές που προέρχονται για από αυτές τις επιδράσεις. Ε, όλα τα κράτη-μέλη επηρεάζονται, αλλά ως τώρα δεν είχαν αναλάβει κοινή δράση. Χαίρομαι που αυτή τη στιγμή, έστω και καθυστερημένα, ε, διαθέτουμε μια νομοθετική πράξη που αναφέρεται στις απειλές των χωροκατακτητικών ξενονιδών. Είναι μάλιστα η πρώτη πρόταση σε 20 χρόνια ε, που αναφέρεται στην ε, μείωση της βιοπικιλίας. Η Κομισιόν προτείνει ένα σχέδιο δράσης για να, να προλάβουμε, ε, να περιορίσουμε ή να μειώσουμε τις ζημιές που μπορούν να προκύψουν από αυτά τα ξένα είδη από την μεταφορά, εξάπλωση και απελευθέρωση αυτών των ειδών. Η Κομισιόν προτείνει ένα σύστημα έγκαιρης απόκρισης. Ε, μία από τις προτάσεις της Κομισιόν αφορά την ε, τεχνολογική ε, υποστήριξη που είναι πολύ σημαντική. Είμαστε σε συνεχή επαφή με την ε, Κομισιόν. Είναι πολύ δημιουργική η προσέγγιση της ως τώρα. Είμαστε γενικά υπέρ των προτάσεων της Κομισιόν. Είναι καλή βάση. Συμφωνώ με την Κομισιόν ότι θα πρέπει να βασιστούμε στην αρχή της πρόληψης, ιεράρχησης και συντονισμού. Απλώς σε ορισμένε περιπτώσεις θα ήταν καλό να ενισχύσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Το βασικό τμήμα της πρότασης προφανώς είναι ο κατάλογος των ειδών στα οποία αναφέρεται. Θα πρέπει να εστιαστούμε λοιπόν στα κριτήρια προετοιμασίας αυτού του καταλόγου. Εγώ εστιάστηκα και σε κάποιε άλλε ανησυχίε, για παράδειγμα, ο κατάλογο αυτό θα πρέπει να συντάσσεται με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Δεύτερον, η Κομισιόν δεν αναφέρεται σε ορισμένα είδη τα οποία εγώ θεωρώ σημαντικά τα οποία δημιουργούν κινδύνους σε κράτη-μέλη, σε πολλά κράτη-μέλη και τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με συνεργασία. Ε, τρίτον, το πρόβλημα είναι ο περιορισμός του καταλόγου σε 50 είδη. Έχω υποβάλει λοιπόν συγκεκριμένες τροπολογίες, πιο συγκεκριμένα τις εξής προτείνω, να αρθεί το όριο των 50 ειδών που θα συμπεριφθούν στο κατάλογο. Για ποιο λόγο. Γιατί, ο λόγος περιγράφεται στην ίδια την μελέτη ε, επιπτώσεων της πρότασης Κομισιόν. Γιατί λέει η Κομισιόν είναι αδύνατο να ξέρουμε εκ των προτέρων ε, ποια και πόσα είδη θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των ε, ε ξένων ειδών. Αυτός είναι ο λόγος. Προτείνω ο κατάλογος αυτός να ε, δημιουργείται με ε, κατεξοδότηση πράξη και όχι εκτελεστικές πράξεις. Θα μπορούσαμε βέβαια να ε, δούμε την ισορροπία ανάμεσα στη λειτουργικότητα και τη δημοκρατικότητα. Εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα χωρίς την συνεργασία όλων και η δημοκρατική αντιμετώπιση θα μας βοηθήσει σε αυτό. Ο κατάλογος θα πρέπει να είναι παράρτημα της βασικής πράξης διότι είναι πολιτικά πολύ σημαντικός και συνδέεται με το πεδίο εφαρμογή της πράξης. Ε, υπάρχει και το θέμα ε, ηθαγενών, ε, ε, ειδών που είναι ηθαγενείς σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης, αλλά ε, σε άλλα. Εδώ ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί ε, ο κατάλογος και με είδη τα οποία είναι ε, προβληματικά για ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν και όχι για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να εξαιρούνται για διοικητικούς λόγους. Επίσης, κάποιες ε, προτάσεις για είδη που είναι ενεφρόντα σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη μπορούν να πάρουν ε, αυστηρότερα μέτρα για αυτά. Αυτό για να ικανοποιήσουμε ε, τα κράτη-μέλη τα οποία ήδη είναι δραστήρια θα πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη λάβει ακόμα και ένα αυστηρότερα από αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Επίσης, χρειαζόμαστε κάποιες αποκλήσεις για να ενισχύσουμε την ε, μελλοντική συμμόρφωση των κρατών μελών με συγκεκριμένες, μέσω συγκεκριμένων ε, αξώνων προτεραιότητας και περιφερειακής ελαστικότητας. Όμως, αυτές οι αποκλήσεις ε, προτείνονται για να ενισχύσουμε την πρόταση της Κομισιόν, όχι για να την αποδυναμώσουμε. Επίσης, ε, πιστεύω θα πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα πληροφοριακή υποστήριξη προτείνει η Κομισιόν και πολύ καλά κάνει, γιατί είναι σημαντικό τμήμα τη ε, πρόταση. Ε, είναι αναπόφευκτο να ενισχυθεί και η συμμετοχή του κοινού. Είναι πολύ κρίσιμη για να πετύχουμε πρόοδο στην καταπολέμηση των χωρακτητικών ξένων ειδών. Θα πρέπει να δούμε σε ποιο επίπεδο όμως. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο το συζητήσαμε αυτό με τους κοιόδες και θα συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Επίσης πρότεινα να δημιουργηθεί ένα ε, ειδικό επιστημονικό φόρουμ για να υποστηρίξει την διαδικασία λήψη αποφάσεις. Ε, το εύρος της απόφασης είναι πολύ πλατή, ε, αυτά τα ξένα είδη είναι πολύ διαφορετικά από τα ε, θηλαστικά ε, ή από τα πουλιά για να μην πούμε διαφορετικά από η θαλάσσια είδη ή μικροοργανισμούς που είναι πραγματικά πολύ μακριά βιολογικά. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε τη γνώμη των επιστημόνων. Δύο πράγματα δεν συμπεριέλαβα στην έκθεσή μου και ελπίζω ότι θα το κάνουμε όλοι μαζί στις επόμενες ε, συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Για παράδειγμα, το ένα θέμα είναι η χρηματοδότηση. Η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι πολύ σαφής. Δεν έχω προτείνει, δεν προτείνω καμία αλλαγή αυτή τη στιγμή στην έκθεσή μου. Θα το συζητήσουμε. Όπως επίσης θα συζητήσουμε και το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων. Υπάρχει ήδη στην έκθεση της Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί. Το συζητήσαμε στην τελευταία συνάντηση των σκιωδών και θα συνεχίσουμε να το συζητάμε και στο μέλλον. Ε, Ω τώρα έχουν λάβει χώρα δύο συναντήσει με του και ηγητέ. Θέλω να του ευχαριστήσω για τα πολύτιμα σχόλιά του. Ε, η συνεργασία είναι πολύ στενή, πολύ καλή, θετική, επικοδομητική Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου και όλους αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκα. Για μένα είναι προσωπικό θέμα. Ε, εγώ εργάστηκα ε, για 20 χρόνια ε, για αυτό το θέμα στη χώρα μου και ζητώ συγγνώμη που μερικές φορές είμαι υπερβολικά ε, συγκεκριμένος. Ε, ε, ελπίζω θα συνεχίσουμε την καλή μας συνεργασία και τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Την κυρία Ζόμερ ποιος την εκπροσωπεί. Ο κύριος Ζέμπερ. Τον ακούμε. Ευχαριστώ. Ε, ζητά συγγνώμη η κυρία Ζόμερ γιατί είχε άλλη υποχρέωση που δεν μπορούσε να την αναβάλει. Εξ ονόματός της λοιπόν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μποκ γιατί ε, πραγματικά έκανε πολύ καλή δουλειά ε, και η συνεργασία του ήταν πολύ καλή. Λίγα είναι τα προβλήματα με την πρότασή του. Γενικώ μπορεί να την υποστηρίξει η κυρία κυρίω κυρίως ό,τι αφορά την συγκέντρωση στα προληπτικά μέτρα που έχουν ως στόχο να προστατεύσουν τη βιοπικιλότητα και να μειώσουν τις ε, συνέπειες στην οικονομία και στην κοινωνία. Ε, νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι σημαντικό. Επίσης, αυτό η θέση των προτεραιοτήτων ε, πρέπει να μιλούσουμε για συγκεκριμένα χωροκατακτητικά είδη και Βέβαια, αυτά τα είδη σε κάποια μέρη της Ευένωσης είναι χωροκατακτητικά, σε, άλλες, σε άλλα μέρη όχι. Ε, βέβαια νομίζω ότι μπορούμε να το, έτσι όπω το προτείνει ο κύριο Ποκ, μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Επίση, ένα ευρωπαϊκό συντονισμό ναι, είναι απαραίτητο έτσι ώστε τα, ε, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων και ε, να χρησιμοποιήσουμε τι συνέργειες που υπάρχουν ε, ή που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ας πούμε, ε, το stop στα όρια του, ε, των συνόρων. Ε, θα πρέπει εδώ να προχωρήσουμε μαζί. Η συμμετοχή επίσης του κοινού είναι πολύ σημαντικό θέμα, κυρίως σε ό,τι αφορά την χρήση των νέων τεχνολογιών. Όλα αυτά τα συμπεριλαμβάνει ο κύριος Πόξ στην έκθεσή του, οπότε τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που έκανε και την πολύ καλή συνεργασία. Το μόνο ένα σημείο που θέλουμε να συζητηθεί είναι αυτή η συμπερίληψη των φυτών που είναι τροποποιη... γενετικώς τροποποιημένα. Ε, αν αυτό ταιριάζει σε αυτή την έκθεση δεν ξέρω, ε, πρέπει να το συζητήσουμε στην ομάδα, ε, ήθελα απλώς να το αναφέρω και να δούμε αν μπορούμε αυτή την ε, πρόταση να την, ε, να την ε, κυρίως, στη, να στοχοθετήσουμε συγγνώμη, στην, στα χωροκατακτητικά η Δεν θέλω βεβαίως να αφήσουμε κατά μέρος τους γενετικώς τροπιωμένους οργανισμούς, απλώς δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζουν αυτοί εδώ, σε αυτή την έκθεση. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια συζήτηση ως προς αυτό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται το σημείο αυτό στην έκθεση, αλλά κατά τα λοιπά συγχαρητήρια για την εξαιρετική σας έκθεση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν ε, μιλάμε για βιοπικιλότητα, φύση, κατά κάποιο τρόπο τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλοί άλλοι φαίνεται να αρχίζουν να παίζουν ε, ένα κρυφτούλι. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε δει επιστημονικές μελέτες ε, για τις ε, τεράστιες ε, ζημιές λόγω των χωροκατακτικών ξένων ειδών. 12 δισεκατομμύρια ευρώ λένε οι μελέτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ζημιά αν ε, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε οικονομικός τομέας είχε τέτοιου επίπεδου ε, απώλειες, θα βλέπατε πολύ σοβαρότερη δράση. Όσον αφορά τα ξένα είδη, οι βασικότεροι κίνδυνοι ε, αφορούν την βιοπικιλότητα. Είτε πρέπει να κάνουμε μια επιλογή, είτε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ισχυρή δράση ή θα πούμε ότι δεν είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν ακούμε την επιστήμη και δεν κάνουμε τίποτα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιλέξει αυτό το 3%, 3% 50 μόνο ήδη, είναι σαν να μην κάνει τίποτα. 3% ή 50 είδη από χιλιάδες ε, χωροκατακτητικά ξένα είδη που είναι υπεύθυνα για 12 δισεκατομμύρια ε, ευρώ σε απώλειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν κανεί στρατηγική της βιοπικιλότητας, ε, τις δεσμεύσεις τις οποίες αναλάβαμε στους στόχους ΑΕΚΙ, υπάρχουν επαρκείς λόγοι να είμαστε πάρα πολύ σοβαρή ω προς την αντιμετώπιση του προβλήματος των χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Οπότε το ερώτημα μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι για ποιο λόγο ε, υποβάλλεται μια τόσο αδύναμη πρόταση. Επιλέγεται 50 ήδη μόνο, ε, δεν μπορώ να την πάρω πολύ σοβαρά. Μπορούμε να την ε, τροποποιήσουμε. Το είπε και ο εισηγητής ότι θέλει να, την, να αλλάξει το 50 ως όριο ειδών. Έχουμε όμως καμιά ιδέα κατά πόσο το, τα κράτη-μέλη έχουν σκοπό να πάρουν σοβαρά αυτό το θέμα ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έλαβε ήδη υπόψη και δεν ακολούθησε την ίδια την, ε, τις ίδιες επιστημονικές μελέτες τις δικές της και αποφάσισε να ακολουθήσει την πολιτική, όχι ηγεσία, αλλά τέλο πάντων ε, κατεύθυνση των κρατών μελών. Εμένα πάρα πολύ με ανησυχεί αυτό το θέμα και πού μπορούμε να φτάσουμε, γιατί με μια τόσο αδύνατη πρόταση ως βάση και μια πιθανή, μια πιθανή αρνητική άποψη κάποιων κρατών μελών μπορεί να μην καταστεί πιθανό να κάνουμε κάτι. όχι μόνο τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ που χάνονται, αλλά και για τις τεράστιες απώλειες βιοπικιλότητας που για, τις, για, για την οποία είναι υπεύθυνα τα χωροκατακτικά ξένα είδη. Όσον αφορά αυτά που είπε ο Πάβελ για την ε, αντιμετώπιση του καταλόγου των 50 ειδών, συμφωνώ απολύτως, είναι κάτι το οποίο πρέπει να πολεμήσουμε. Κάτι ακόμη που θα ήθελα να προσθέσω είναι να συμπεριλάβουμε επίσης το θέμα της ασφάλειας. Στη δική μου χώρα, στις κάτω χώρες, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με ένα είδος ε, ποντικού που βρίσκεται κάτω από τα ορυχεία. Είναι πράγματι ένα χωροκατακτητικό ξένο είδος και πρέπει πραγματικά να το καταπολεμήσουμε για να σώσουμε από τις πλημμύρες ε, τις ε, κάτω χώρες. Ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες με το ζώο αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τα τρόφιμα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στον τομέα της γεωργίας με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Οπότε η έκκλησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρακαλώ λάβετε υπόψη, μου, υπόψη σας την έκκληση προς τα κράτη-μέλη όταν το συζητάτε μαζί τους, ε, πάρτε το σοβαρά και μην σκέφτεστε ότι αφορούν μόνο το θέμα, αφορά μόνο το θέμα της βιοπικιλότητας και της φύσης ε, και να συνεχιστεί αυτό το κρυφτούλι ε, και να κάνουμε στον σε σχέση με τις αποδείξεις που μας παρέχουν τα επιστημονικά στοιχεία. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ ισχυρή έκθεση. Η έκθεση του Πάβελ νομίζω ότι είναι ε, ήδη πολύ ε, ισχυρή στον τόνο της, ε, πολύ έντονη στον τόνο της και πιστεύω ότι θα είναι πολύ ισχυρή και η θέση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Πολύ λέει ο κύριος Ντέμες Μέκερ. επιτέλους επιτέλους αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να συμφωνήσω απολύτως με όσους έλαβαν το λόγο πριν από μένα. Πολλά χρόνια υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, μια μεγάλη απειλή για τη βιοπικιλότητα. Στο φλαμαντικό Κοινοβούλιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο εγώ προσπάθησα τέτοιου είδους διατάξεις ε, να εγκριθούν, συχνά η δράση είναι τόσο κατακαιρματισμένη που δεν είναι πια αποτελεσματική. Τα χωροκτακτητικά είδη, ε, ξένα είδη, ε, δεν γνωρίζουν σύνορα και είναι ένα από τα συγκεκριμένα παραδείγματα που μας δείχνουν πόσο ένας ευρωπαϊκός συντονισμός θα μπορούσε να επιφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία. Ως σκιώδης εισηγητής των Πρασίνων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Πάβελ Ποκ ε, για τη μέθοδο εργασίας του που είναι πάρα πολύ επικοδομητική. Να τον συγχαρώ επίσης ε, για την πρακτική προσέγγιση του. Νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά η καλύτερη λύση και η πιο αποτελεσματική. Επίσης, ε, να συγχαρώ σε σχέση με το αυθαίρετο του ανώτατου ορίου των 50 ειδών και την περίοδο την πενταετή που προβλέπεται στο άρθρο 19. Να συγχαρώ τον εισηγητή λοιπόν για αυτά που λέει σε σχέση με τα θέματα αυτά. Είναι πολύ σύντομη αυτή η περίοδος για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Μήπως μπορούμε να πάμε λίγο πιο πέρα από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει ποιες είναι αυτές οι πιθανότητες να πάμε λίγο πιο πέρα. Και επίσης η συμμετοχή σε ένα επιστημονικό φόρουμ των επιστημόνων. Ναι, αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Ζητήσαμε διευκρινήσεις. Οι διατάξεις που μας δημιουργούν πρόβλημα είναι οι 4 και οι 24 προβλέπουν ένα σύστημα παρέκκληση σε εθνικό επίπεδο εγώ δεν θα ήθελα να υπάρχει δυνατότητα ad hoc δράσεων που μπορούν να αποδυναμώσουν μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει αναστάτωση στις αγορές. Κάτι ακόμη γιατί θα υποβάλω εγώ τροπολογίες. Όσον αφορά την καταπολέμηση των ειδών αυτών, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ευαισθητοποίηση ε, του πληθυσμού, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα θέματα ευημερία των ζώων και δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει ένα σύστημα ελέγχου θα έπρεπε να βασίζεται σε καλούς ελέγχους στα κρατημέλη και τρίτον, είναι ουσιώδες από απόψεως χρηματοδότησης και προϋπολογισμού για τα μέτρα αυτά να κάνουμε όλον τον απαραίτητο σχεδιασμό και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει ήδη το αυριανό εργαστήριο περιμέναμε για καιρό αυτή την ε, πρόταση και αυτό οφείλεται όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις στο ότι η Κομισιόν συμφωνούσε εσωτερικά για την πρόταση. Βλέποντας την πρόταση μάλιστα βλέπουμε ότι δεν είναι και πολύ φιλόδοξη. Ε, όμως ε, με την βοήθεια του κ. Ποκ που καταλαβαίνει την, το θέμα ε, μπορούμε ε, να βελτιώσουμε αυτή την πρόταση σε συνεργασία, σε εργαστή συνεργασία μέχρι τώρα. Ε, νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό παρανομαστή μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων. Όλα τα κράτη-μέρη άλλωστε παίρνουν πολύ στα σοβαρά αυτό το θέμα. Βέβαια έχουν άλλες προσεγγίσεις. 12 κράτη-μέλη επιβάλλουν εισαγωγικούς περιορισμούς. 11 ε, με κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τέσσερις διαφορετικές μεθόδους ε, αξιολόγησης του κινδύνου. Δεν προτείνω συχνά εναρμόνιση, αλλά σε αυτόν τον τομέα νομίζω είναι πολύ σημαντικό όλοι να εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση και με τον ίδιο στόχο. Ακροθυγώς αναφέρθηκε ε, το γεγονός ότι ε, μπορεί ε, το να μην έχουμε ε, να μας υποστηρίξει εύκολα κοινή γνώμη, γι' αυτό λόγο πρέπει να έχουμε σοβαρά και ισχυρά επιχειρήματα. Υποστηρίζω και εγώ λοιπόν τον εισηγητή που προτείνει την κατάργηση αυτού του ανώτατου ορίου των 50 ειδών. Κανένας δεν το υποστηρίζει αυτό. Ούτε και τα κράτη-μέλη πιστεύω στο Συμβούλιο. Οπότε ελπίζω ότι γι' αυτό και για κάποια άλλα πράγματα θα συμφωνήσουμε πολύ γρήγορα. Ε, οι θαγενή ήδη που είναι χωροκατακτικά σε άλλη χώρα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Ε, τα κράτη-μέλη θα μπορούν επίσης να λαμβάνουν πιο αυστηρά μέτρα όπου χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά με έλεγχο. Με έλεγχο. Επιπλέον μπορεί να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τις παρεκκλήσεις. Όχι πως δεν θα έπρεπε να προβλέψουμε μηχανισμό παρέκκλησης θα έπρεπε, αλλά με ανησυχεί το ότι οι εθνικές αποκλήσεις όπως προτείνονται από τον εισηγητή μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δηλαδή είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν ως παραθυράκι για τη μη εφαρμογή των κανόνων. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε τις παρεκκλήσεις έτσι ώστε να μην πληγεί ο τελικός στόχος. Ε, κατόπιν, για το θέμα των γενετικά τροπημένων οργανισμών, θα ήταν επικίνδυνο, πιστεύω, να επιτρέψουμε αυτή η έκθεση να παρεκτραπεί σε μια συζήτηση των, ε, του θέματος ε, των γενετικά τροπημένων οργανισμών. Θα ήταν λάθος πραγματικά να εισάγουμε το θέμα των γενετικά τροπημένων οργανισμών σε αυτή την έκθεση. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πόλωση σχετικά με τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς και δεν θα ήθελα ε, το θέμα αυτό να καθυστερήσει ε, ή να αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης εξαιτία της αναφοράς σε γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Ας τους αφήσουμε εκτός λοιπόν. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ja, dank u wel. Allereerst zou ik de rapporteur, de heer hartelijk willen bedanken. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και εγώ για την πρότασή του, για τη συνεργασία που είχε με τους σκιώδες. Δεν έχω πολλά να προσθέσω στα όσα είπαν οι συνάδελφοι σκιώδες εισηγητές. Απλώς ε, κάποια σημεία θα ήθελα να σχολιάσω. Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή. Δεν χρειαζόμαστε αυτό το όριο των 50 ειδών. Αυτό θα πρέπει όντως να βγει από την έκθεση. Και αν μιλούμε για 1.200 ή 1.400 κατακτητικά είδη, ε, προφανώς δεν μπορούμε να βρούμε τα 50 και να τους δώσουμε διακριτική μεταχείριση. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί σε ό,τι αφορά την αρχή της πρόληψης, θα πρέπει να προχωρήσουμε όντως προληπτικά και όχι να επικεντρωθούμε μόνο σε αυτά τα 50 είδη, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να αναπτύσσονται ελεύθερα. Επίσης, το θέμα της βιοπικιλότητας. Ναι, πρέπει να προστατεύσουμε την ε, βιοπικιλότητα προφανώς. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να αποφύγουμε αρκετά μεγάλα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν για τα ζώα. Η Κομισιόν βεβαίως δεν μιλάει για την ευζοία των ζώων, όταν μιλούμε για χωροκτητικά ξένα είδη, τότε είναι σαφές ότι υπάρχουν αρκετά είδη ζώων, τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ο πιο γρήγορος ε, α, τρόπος ε, βέβαια είναι να τα θανατώσουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι η τελευταία μας επιλογή. Αν ξεκινήσουμε τώρα τη θανάτωση, ε, τότε ε, θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο φιλική προς το ζώο αυτή η επιλογή. Δεν μπορούμε έτσι να πάμε απλά και να τα σκοτώσουμε. Κάποιοι συνάδελφοι μίλησαν για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και είπαν ότι πρέπει να αποκλειστούν από την ε, έκθεση αυτή, να μην μπουν στο πεδίο εφαρμογή. Αλλά αν δείτε του ορισμού στην πρόταση τη Κομισιόν, δεν θέλω τώρα να μπω σε όλε τι λεπτομέρειε, αλλά μιλάει για τα χωροκατακτητικά είδη και η εισαγωγή λέει ε, απειλούν τη βιοπικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Ε, νομίζω ότι αυτό ο ορισμό ισχύει για τους γενετικώ οργανισμούς, γιατί τα φυτά ας πούμε, που είναι γενετικώς τροποποιημένα μπορεί να αποτελέσουν ένα είδος μόλυνσης, μπορεί να κατακτήσουν άλλα φυτά. Οπότε νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μείνουν εκτός οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί, γιατί ταιριάζουν με αυτόν τον ορισμό. Και επίσης συμφωνώ με τον εισηγητή ότι αν υπάρχουν κρατημέλη που θέλουν να λάβουν πιο αυστηρά μέτρα, ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό γίνεται. Και βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει η σωστή πληροφόρηση προ το ε, κοινό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριο κύριος Μπάνκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ μιλούμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όντως είναι ιδιαίτερα σοβαρό Υπάρχουν διάφορα ε, φυτά τα οποία προκαλούν αλλεργίες σε διάφορα κρατημέλη και αυτά τα φυτά είναι ιδιαίτερως διαδεδομένα. Τέτοια φυτά υπάρχουν και στην ε, Ουγγαρία. Με την ε, πρόταση το πρόβλημα είναι το εξής. Ορίζεται, μάλλον διαπιστώνεται ότι οι ζημίες λόγω αυτών των ειδών για τα οποία μιλούμε φτάνουν τα 12, τα 12 Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, αυτές οι ζημίες που προκαλούνται φτάνουν περίπου τα 200.000 ευρώ. Βεβαίως αυτό αφορά ένα είδος μονάχα. Ε, και επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κάθε χώρα που βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε πιο δύσκολη θέση από τις υπόλοιπες. Ακόμη και αν δημιουργήσουμε λοιπόν μία διάταξη που θα λέει τι γίνεται σε περίπτωση τέτοιων, ύπαρξης τέτοιων χωροκατακτητικών ειδών, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης θα έχουν πιο μεγάλες δυσκολίες να την εφαρμόσουν, γιατί προφανώς ε, ε, εκτίθενται σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτά τα είδη. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια κοινή στρατηγική, ένας κοινός μηχανισμός, στον, ε, στην χρηματοδότηση του οποίου θα συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω, θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή στρατηγική η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τα διάφορα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητε τη ε, κάθε χώρα. Επίση, εξίσου σημαντικό είναι όταν μιλούμε για το ευρωπαϊκό επίπεδο και αν θέλουμε να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, κυρίως για αυτά τα χωροκρατητικά είδη, και αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες ασθένειες, τις διάφορες αλλεργίες που προκαλούνται από αυτά τα είδη, αν θέλουμε να μειώσουμε τις ζημίες που προκαλούν αυτά τα είδη, τότε θα πρέπει να δράσουμε μαζί. Αλλά αυτή η κοινή δράση δεν θα πρέπει να αποτελείται μόνο από υποχρεώσεις, θα πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα κονδύλια, τα απαραίτητα μέσα για να γίνουν όλα αυτά. έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουν και στη λύση των προβλημάτων των διαφόρων κρατών μελών, τα οποία βεβαίω ε, εκτίθενται σε πολύ διαφορετικό βαθμό σε αυτά τα προβλήματα και σε αυτά τα είδη και προφανώς χρειάζονται και διαφορετικές στρατηγικές. Ευχαριστώ να ακούσουμε την, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Thank you, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο σήμερα και θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως ιδιαίτερα τον ε, εισηγητή τον Παύλ Ποκ για την πολύ διεξοδική εργασία του που είναι και εξαιρετική ως τώρα σε σχέση με την πρότασή μας. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω όλους ε, για την ε, πραγματική αφοσίωση που δείχνεται στο στόχο της ε, προσπάθειες ολοκλήρωσης αυτού του θέματος πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε άλλωστε όλοι, είναι ένα θέμα που ανησυχεί όλους μας και όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, να σας εξηγήσω τη λογική της πρότασής μας, ε, η οποία μπορεί να λύσει και κάποια προβλήματα που ε, είχατε σε σχέση με την ε, πρότασή μας και να διασκεδάσει κάποιες ανησυχίες. Είδαμε το θέμα της αρχής επικουρικότητας. Υπάρχει ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να παρέμβουμε όταν ε, θα υπάρξει προστιθέμενη αξία από πλευράς Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης αν η δράση είναι ευρωπαϊκού επίπεδου, όταν μπορεί να αφαιθεί ε, σε εθνικά χέρια η δράση είναι καλύτερα να ε, γίνει αυτό. Είναι καλύτερα να αναλυφθεί δράση σε επίπεδο κρατών μελών. Γι' αυτό ακριβώς προτείναμε, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την πρότασή της και οι δύο συνομοθέτες ε, θα πάρουν τις αποφάσεις τους, γι' αυτό λοιπόν προτείναμε να ε, ασχοληθούμε μόνο με είδη τα οποία ανησυχούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και γι' αυτό προτείναμε αυτόν τον αριθμό των ε, χωροκατακτητικών ξένων ειδών που αφορούν ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς υπάρχουν κάποια είδη τα οποία ε, είναι αντικείμενο δράσης σε επίπεδο ε, κρατών μελών και υπάρχουν και είδη τα οποία απασχολούν σε περιφερειακό επίπεδο κάποια κρατημέλη αλλά όχι κάποια άλλα. Και γι' αυτό η άποψή μας ήταν ότι θα ήταν καλύτερο σε πρώτη φάση να ασχοληθούμε καλύτερα με αυτά τα είδη που αφορούν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αφήσουμε στα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο βέβαια των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, τη μέρημνα να ε, προχωρήσουν ε, στην αντιμετώπιση θεμάτων ε, εθνικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας. Να επανέλθω τώρα σε ορισμένα ζητήματα που ετέθησαν όσον αφορά το ανώδατο όριο που προτάθηκε, ο αριθμός των 50 ειδών. Νομίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο το οποίο ήταν αντικείμενο σχεδόν ομόφωνης απόφασης, ε, αντίδρασης και σε επίπεδο κοινοβουλίου αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Έγινε συζήτηση στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος την Παρασκευή και εκτός από ένα ή κρατημέλη όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη συμφωνούσαν ε, σε γενικές γραμμές με τις απόψεις τις δικές σας που άκουσα σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει και εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσουμε ξανά την πρότασή μας, να ακούσουμε και τη δική σας άποψη και των κρατών μελών. Να σας εξηγήσω λοιπόν γιατί προτείναμε τόσο περιορισμένο αριθμό ειδών. Νομίζω ότι ο κύριος Χερπράντ ρώτησε ποια ήταν η λογική πίσω από την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποιο ήταν το σκεπτικό μας. Το σκεπτικό μας ήταν να μην υπερφορτώσουμε το μηχανισμό από την αρχή. Το σκεπτικό μας ήταν να εξασφαλίσουμε ότι καταρχάς θα μπορούσαμε να αρχίσουμε τη δουλειά και μάλιστα να την αρχίσουμε σε, επιστημονική βάση, σε ορθή βάση και γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε ότι θα ήταν ασφαλές να προτείνουμε ένα νότατο όριο. Βέβαια, όπως είπα, ακούσαμε σχόλια και από τα κρατη και από εσάς σήμερα και θα συνεργαστούμε με όλους σας προκειμένου να βρεθεί μια λύση που ε, θα είναι αποδεκτή για όλους. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο θέμα των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Το θέμα αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει όλους τους νομοθέτες ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ενδιαφέρει και πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες. Όλοι έχουν μία άποψη για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και επειδή είναι σημαντικό θέμα, φρονούμε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε οριζόντιο επίπεδο και πιστεύουμε επίσης ότι ένα τόσο τεχνικό νομοθέτημα δεν θα ήταν, ε, ένα, δεν θα το κατάλληλο θέμα για να αρχίσει βάσει αυτού ε, ένας ολόκληρος πόλεμος για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Γι' αυτό ακριβώς εγώ προσωπικά θα συμβουλέψω ε, τους ανωτέρους μου να επιμείνουν στην πρόταση ότι οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί θα, δεν θα έπρεπε να αποτελέσουν τμήμα του κανονισμού αυτού ως προς την ανάγκη συμπερίληψης όλων των εμπλεκομένων φορέων, των πολιτών, του Εβραίου κοινού. Υπάρχει μία παράθεση από τη Σύμβαση Άρχους για την εξασφάλιση της δημόσιας ενημέρωσης και της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έχουμε νομοθεσία ad hoc σε ευρωπαϊκό επίπεδο που μεταγράφει την σύμβαση του Άρχουσος προς αυτό το θέμα και πρέπει να εξασφαλίσουμε βεβαίως ότι το κοινό συμμετέχει σωστά στην ε, αντιμετώπιση του θέματος των χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Όσον αφορά το θέμα των ε, παρεκκλήσεων, των εξαιρέσεων. Υπάρχουν πολλά αιτήματα αντιμετώπιση του θέματος των εξαιρέσεων υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες. Εμείς προτείναμε να κάνουμε αξιολόγηση κινδύνου, που αυτή η αξιολόγηση κινδύνου βέβαια θα είναι η βάση για το κατά πόσο θα προταθεί να συμπεριληφθεί ένα είδος ή όχι στον κατάλογο. Ο, η αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει να λάβει υπόψη την επιστημονική σημασία της ζημιάς, το γεγονός ότι είναι ξένο είδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση το είδος αυτό, αλλά επίσης εκτός από το ότι είναι ξένο δημιουργεί και πρόβλημα, έχει επιβλαβή επίπτωση και πρέπει να δούμε επίσης και το θέμα της αναλογικότητας, της εξάλληψης του είδους σε σχέση με τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία είναι ήδη επιβεβαιωμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο προσπαθήσαμε να σταθμίσουμε πολύ προσεκτικά πριν ε, διατυπώσουμε τα κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου γιατί αναγνωρίζουμε πλήρως ότι κάποια είδη τα οποία είναι de facto χωροκατακτητικά και ξένα είναι περιορισμένα, είναι σε περιορισμένα ε, περιβάλλοντα ε, στο πλαίσιο των κρατών μελών ε, και έχουν βέβαια και κάποια σημαντική οικονομική αξία. Και γι' αυτό το λόγο η αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να λαμβάνει υπόψη δεόντως και την οικονομική σημασία του είδους, ώστε να μπορούμε να εξισορροπήσουμε και τα δύο στοιχεία. Πρέπει να δούμε και την προστασία, τη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Και γι' αυτό δεν μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη μόνο τη βιοπικιλότητα χωρίς να λάβουμε υπόψη το θέμα της αηφόρου ανάπτυξης γενικότερα και βεβαίως χωρίς να λάβουμε υπόψη το θέμα της ε, ε, προοπτικής, ε, της οικονομικής και τι επίπτωση έχει βέβαια στις θέσεις απασχόλησης. Όσον αφορά ε, τα είδη που δεν είναι ηθαγενή σε, ε, σε συγκεκριμένο κράτος μέλος ή την περιφερειακή διάσταση κάποιων χωροκατακτητικών ειδών, α, ως προς αυτό ανέφερα ήδη πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να επαφίεται στην επικουρικότητα. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα κύριε Πρόεδρε. Είμαστε βεβαίως στη διάθεσή σας και στη διάθεση του εισηγητή και στη διάθεση όλων των υπολείπων ευρωβουλευτών, ε, μελών της Επιτροπής σας, για να συνεργαστούμε μαζί σας, να εξετάσουμε περαιτέρω το ζήτημα και αναμένουμε εναγωνίως συνέχιση της ε, τρέχουσας εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε στον εισηγητή το λόγο. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες όσους πήραν το λόγο για την υποστήριξή τους. Είναι τιμή για μένα. Μερικές παρατηρήσεις για τις κάποιες ανησυχίες που εκφράστηκαν. Μη, ε, γενετικά τροπημένοι οργανισμοί. Φαίνεται ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα. έκπληξη, ε. Πρέπει να συζητηθεί. Και χαίρομαι που η κυρία Σόμερ ε, προτάθηκε από το ΕΛΚΟ συσυγήτρια και θα με βοηθήσει, γνωρίζει πολύ καλά τα γεωργικά. Είμαι ανοιχτό να το συζητήσουμε. Uh, uh, παρεκκλήσεις. Οι παρεκκλήσεις αυτές δεν προτείνονται για να αποδυναμωθεί το κείμενο της Κομισιόν. έχω διαπραγματευτεί για 20 χρόνια με τις τοπικές κυβερνήσεις και η εμπειρία μου δείχνει ότι για στην καταπολέμηση των χωρακατακτητικών ξένων ε, για να πετύχουμε χρειάζεται να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση και η νομοθεσία που προτείνουμε θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για με, τη μελλοντική επιτυχία των προτάσεων. σε ό,τι αφορά τη γνώμη των κρατών μελών. Ε, το έχω συζητήσει το θέμα με πολλούς εκπροσώπους των κρατών μελών στην Κοινή Επιτροπή Γεωργίας. Στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, συγγνώμη. Και νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε καλή συνένεση. Ευχαριστώ τον κύριο Κεμπράντη για την παρατήρηση του περί ασφαλείας. Ε, ελπίζω να μπορέσουμε να το συμπεριλάβουμε Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες, την τελευταία παρατήρηση περί ηθαγενών σε, ένα, σε μια περιοχή ειδών που είναι χωροκατακτητικά σε άλλες περιοχές. Ε, μπορούμε ασφαλώς να το συζητήσουμε με την Κομισιόν. και αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν από πέντε είδη τα οποία εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και μετά θα δούμε αν είναι θέμα επικορικότητας ή θέμα ευρωπαϊκής σημασίας. Θα ήθελα να σας καλέσω αύριο στην συζήτηση θα γίνει για τα χωρακτηριστικά ξένα είδη. Εν πάση περιπτώσει, σα ευχαριστώ όλους. Yeah, that's Vielen Dank, Ευχαριστούμε Πάβελ για τη δουλειά που έκανες, για τη δέσμευση που έδειξες στο θέμα αυτό. Προθεσμία 8 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι για τις της τροπολογίες, 30 Ιανουαρίου εδώ στην Επιτροπή, συζήτηση μαζί με τις τροπολογίες, Επιτροπή Περιβάλλοντος 12-13 Φεβρουαρίου στην, για ψηφοφορία και Ολομέλεια Μαρτίου ή Απριλίου για την ε, τελική ψηφοφορία. Πάμε στο σημείο 12 της σημερινής διάταξης. Ο κύριος Ζέμπερ θα προσωπήσει την εισηγήτρια. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συνάδελφος Αντωνέσκου δεν είναι εδώ, οπότε πρέπει να την ε, εκπροσωπήσω, αλλά επειδή δεν μπορώ να μιλήσω τόσο καλά ε, ε, ρουμανικά, θα διαβάσω το κείμενό της στα αγγλικά. The show must go on, colleagues. <laughs> so, but let's, let's continue in English. Η παράσταση πρέπει να έχει συνεχιστεί, συνάδελφοι. Α συνεχίσω το κείμενο στα αγγλικά. Δεν είναι δυνατόν να είναι εδώ η συνάδελφο. Μου ζήτησε να την αντικαταστήσω και Προετοίμασε το εξή ε, κείμενο. Το 2010 υπέβαλε μία προφορική ερώτηση σε σχέση με τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες. Ε, υπήρξε μεγάλη Μεγαλό διάλογο για το θέμα αυτό σε κάποιες από τις συνεδριάσεις Επιτροπή μας. Επειδή υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, ε, ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πρόθεση έχει σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αυτά τα ε, αυξανόμενα φαινόμενα. Ε, νέα ψυχοτρόπος ουσία σημαίνει μία ουσία η οποία όταν ε, καταναλώνεται από έναν ε, ανθρώπινο οργανισμό υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει παρεστήσεις, αλλαγές στις κινητικές του συνήθειες κλπ επειδή υπάρχει νέο, νέα παρακολούθηση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ναρκωτικών Ουσιών, ε, νέων ψυχοτρόπων ουσιών, αναφέρθηκαν νέες ε, ψυχοτρόπες ουσίες, συγκεκριμένα ε, τριπλασιάστηκαν από 24 σε 73 μέσα σε τρία χρόνια. Ε, πάνω από ένα κράτος μέλος ε, ανέφεραν την αύξηση αυτή. Μπορεί να πάμε και σε χιλιάδες ουσίες γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ε, διαφορετικές ποικιλίε, μπορούν να γίνουν διαφορετικές αλλοιώσεις των ουσιών αυτών, κάτι το οποίο βέβαια μπορεί να είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία και τη δημόσια υγεία, μπορεί ε, να οδηγήσει σε σοβαρές ασθένειες μέχρι και στο θάνατο. Γι' αυτό ακριβώς ε, πολλές τέτοιες ψυχοτρόπες ουσίες είναι επικίνδυνες γιατί πολλούνται χωρίς την απαραίτητη ετικετοθεσία, είναι αντικείμενο εμπορευματοποίησης ε, και αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρξει ένα τρόπο, ένα μηχανισμό ανταλλαγή πληροφοριών νέων ψυχοτρόπων ουσιών που, αναφέρονται, που ε, τοποθετούνται στο εμπόριο για ε, βιομηχανική χρήση, αξιολόγηση των ε, ουσιών αυτών και εξέταση του ενδεχομένου απόσυρση από το εμπόριο των, χωρών που των ουσιών που δημιουργούν πρόβλημα. Πολλά ε, στοιχεία της ε, νέας πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σημαίνουν καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η ραγδαία αυξανόμενη αγορά νέων ψυχοτρόπων ουσιών. Πρόκειται για έναν καλό μηχανισμό, όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα γιατί είναι πολύ χρονοβόρος ο μηχανισμός και δεν υπάρχουν επαρκή ε, μέτρα ε, για τη διενέργεια ελέγχων και για την ύπαρξη κυρώσεων σε περίπτωση εγκληματικών πράξεων. Ε, ειδικότερα για το θέμα των άμεσων κινδύνων για τη δημόσια υγεία, οι σχετικές ουσίες πρέπει να αποσύρονται αμέσως από την αγορά. Αφού γίνει αξιολόγηση κινδύνου, πρέπει να είναι αναλογικά τα μέτρα σε σχέση με την επικινδυνότητα της ουσίας. Ε, δεν θα υπάρξουν όμως ε, αλλαγές σε σχέση με ε, ουσίες που δημιουργούν χαμηλούς ή μέτριους κινδύνους για τη δημόσια υγεία όταν είναι σωστά οριοθετημένη η χρήση τους στην αγορά ή συγκεκριμένα επιτρέπονται στο πλαίσιο μιας ιατρικής νομοθεσία ή για εμπορικούς βιομηχανικούς λόγους ή για ερευνητικούς λόγους οι νέες ψυχοτρόπες ουσίες που δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους θα υπόκεινται σε μόνιμη απαγόρευση από την αγορά και για τους καταναλωτές και ε, για το εμπόριο και η χρήση θα μπορούσε να γίνει μόνο για συγκεκριμένους βιομηχανικούς λόγους ή για ε, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη. Επίσης ε, θα, υπάρξει, θα, υπάρξουν, θα, υπάρχουν, ε, θα υπάρχει ένας μηχανισμός ε, κυρώσεων σε περίπτωση παράνομης διακίνησης και λάθος χρήσης των ουσιών αυτών για να εισαχθούν κάποια στοιχεία τα οποία βέβαια έχουν να κάνουν με την δική μας, με την αρμοδιότητα της δική μας επιτροπή. Ε, ο Οργανισμός ε, Χημικών ε, και Φαρμάκων και Ελέγχου Νόσων θα έπρεπε επίσης να συμμετέχουν όλοι αυτοί οι οργανισμοί στην αξιολόγηση των νέων ψυχοτρόπων ουσιών. Επίσης η συγγήτρια ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις αντενδείξεις με άλλες ουσίες όταν καθαρίζεται το επίπεδο ε, του κινδύνου ε, που υπάρχει ε, λόγω μιας νέας ψυχοτρόπου ουσίας. Σε σχέση με τη διαδικασία ανταλλαγή πληροφοριών του άρθρου 5, πιστεύει ότι οι πληροφορίες των εθνικών σημείων εστίασης και των εθνικών μονάδων της Europol προς τον οργανισμό ε, ελέγχου νόσων και την ίδια τη Europol ε, πρέπει να αφορά τα συγκεκριμένα στοιχεία των νέων ψυχοτροπιών ουσιών και συγκεκριμένες ε, ουσίες και συγκεκριμένα, συγκεκριμένες, συγκεκριμένα ανάμιξη ουσιών που μπορεί να είναι επιβλαβής ή θανατηφόρα για τον ανθρώπινο οργανισμό πιστεύει ότι για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη χρήση των νέων ψυχοτρόπων ουσιών και των ενδεχομένων κινδύνων τους, τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, έχουν προγράμματα πρόληψης και να ευαισθητοποιήσουν ε, τους πολίτες τους σε σχέση με τις συνέπειες χρήσης τέτοιων ουσιών. Όσον αφορά τις ουσίες που δημιουργούν χαμηλό ε, κίνδυνο, προκαλούν χαμηλό κίνδυνο, πιστεύει η ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το είδος αυτών των κινδύνων, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ένα είδος ουσίας μπορεί να προκαλεί χαμηλό κίνδυνο για την υγεία. Ε, πιστεύει ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και να ληφθούν και άλλου είδου υπόψη, άλλου είδου παράγοντες υπόψη όπω ε, οι τάσει κατανάλωση, η συχνότητα χρήση και η σχέση της χρήση παράλληλα με άλλε ουσίες. Και ε, ολοκληρώνοντας, η συγγήτρια θα ήθελε να τονίσει ότι επικροτεί την πρόταση του κανονισμού που είναι κάτι που το περιμέναμε πολύ καιρό το φαινόμενο των νέων ψυχοτρόπων ουσιών είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, εξαιρετικά επικίνδυνο και η συγγήτρια πιστεύει ότι ο κανονισμός αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί, να συμπληρωθεί με δράσεις και μέτρα που θα λάβουν τα κράτη-μέλη. Αναμένει ένα γωνίο συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητής και με τους υπόλοιπους συναδέλφους της Επιτροπής μας, όπως επίσης και με τον κύριο Προτασίεβιτς από την Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Έναν σκιώδη έχουμε εδώ. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Σουσόγγελος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Το ζήτημα του ελέγχου της παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης των νέων ψυχότροπων ουσιών είναι πολύπλοκο και χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση με έμφαση στην πρόληψη, θεραπεία, παρακολούθηση, έγκαιρη αντιμετώπιση μείωση τη βλάβη και βελτίωση του νομικού πλαισίου, καθώ δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση που να ταιριάζει για όλε τι περιπτώσει, ιδιαίτερα αν εμένει στη λογική του ελέγχου διαμέσου τη απαγόρευση και τη αστυνόμευση. Το απαγορευτικό πλαίσιο και οι κατασταλτικέ πολιτικέ για τι ουσίε, ιδιαίτερα για την πιο διαδομένη από αυτέ, την κάναβη, έχουν ω αποτέλεσμα την είσοδο στην αγορά νέων επικίνδυνων ψυχότροπων ουσιών που δεν περιλαμβάνονται στι λίστε ελέγχου και παρουσιάζονται σαν νόμιμα υποκατάστατα των παράνομων ουσιών, ξεφεύγοντα από το γράμμα του νόμου. Ο αριθμός των νέων ψυχοτρόπων ουσιών που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη-μέλη στα Ηνωμένα Έθνη αυξήθηκε κατά 50% από το 2009 μέχρι το 2012, δηλαδή 166 νέες ουσίες το 2009 που έφτασαν τις 251 μέχρι τα μέσα του 2012. Κατά τη διάρκεια μόνο του 2012 τα κράτη-μέλη κοινοποίησαν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για πρώτη φορά 73 νέες ψυχοδραστικές ουσίες, αποτέλεσμα της αδιάκοπης προσπάθειας να ξεφύγουν από το γράμμα του νόμου που τις καθιστά παράνομες και μη ελέγξιμες. Απ' την άλλη, περισσότερες ουσίες που περιλαμβάνονταν στις λύσει των ΗΠΑ από το 1961 και το 1971 δεν υφίστανται πλέον στην αγορά. Από τις 234 που υπόκεινται σε καθιστός ελέγχου, μόνο μία ντουζίνα από αυτές προκαλούν ανησυχία για, τα, για προβληματική χρήση, ενώ η χρήση πολλών από αυτές μειώθηκε δραματικά χωρίς να έχουν κατηγοροποιηθεί ως παράνομες. Η πρώτη επιτροπή εστιάζει στην ταχύτερη αναγνώριση, την εκτίμηση του κινδύνου και την πιθανή απαγόρευση των ουσιών προκαλούν ανησυχία. Η επαρκή αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων βάσει επιστημονικών αποδείξεων είναι φυσικά πολύ σημαντική αλλά όπω έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια, ακόμα και το πιο βελτιωμένο σύστημα αναγνώριση και έγκαιρη προειδοποίηση δεν θα συμβαδίσει με την ταχύ ανάπτυξη των νέων ουσιών και τα πρότυπα χρήση. Ω εκ τούτου θα υπάρχουν πάντα νέε ουσίε που διανέμονται έξω από το σύστημα ελέγχου, ενώ ακολουθούνται κατά γράμμα διαδικασίε. Μπορούμε επίση να υποθέσουμε ότι ορισμένε από τι ουσίε που αξιολογούνται με, οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα θα κριθούν ότι δεν απαιτούν απαγόρευση. Για τις αυτές θα πρέπει ως εκ τούτου να, αναζητηθούν άλλοι μηχανισμοί για την αναζήτηση των πιθανών βλαβών. Οι προτάσει της Επιτροπής δεν αφορούν επί του παρόντο το πολύ πραγματικό φαινόμενο τη μετατόπιση από τη μία ουσία στην άλλη και τη αλλαγή των προτύπων χρήση. Η αύξηση δημοτικότητα των πιο ευρέως δεδομένων νέων ψυχοτρόπων ουσιών τα τελευταία χρόνια είναι τουλάχιστον μέρη αποτέλεσμα των αλλαγών στα πρότυπα χρήση καθώς οι χρήστες απομακρύνονται από ουσίες οι οποίες έχει καταστεί δύσκολη πρόσβαση, π.χ. κάναβη, ή που η ποιότητά τους έχει χειροτερεύσει μέσω της αλλαγής στη δυναμική της αγοράς. Αυτή η γρήγορη αναλλαγή μεταξύ ουσιών που δεν έχει υπολογιστεί ε, ακόμα η βλάβη τους αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ενώ ελοχεύει ο κίνδυνος ένα σύστημα που χτίστηκε αποκλειστικά για τον εντοπισμό και την απαγόρευση συγκεκριμένων ουσιών θα χρησιμεύσει μόνο για να εντείνει αυτή την εναλλαγή στα πρότυπα χρήση. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε οι προτάσει τη Επιτροπή να δώσουν πολύ μεγαλύτερη σημασία σε άλλε μορφέ ελέγχου και προστασία τη δημόσια υγεία, που μα ενδιαφέρει και εμά εδώ ω Επιτροπή, όπω για παράδειγμα η ταχύ αναγνώριση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία ορισμένων ουσιών, π.χ. μέσω του επιτόπου, επιτόπιου ελέγχου και άμεση διάδοση συμβουλών για την προστασία τη δημόσια υγεία και των καταναλωτών η ρύθμιση ορισμένων ουσιών βάσει τη υπάρχουσα νομοθεσία και την προστασία των καταναλωτών ή ακόμα και η δυνατότητα συνεργασία με του πιθανού παραγού για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των καταναλωτών. Σχετικά με το τελευταίο, δεν γίνεται καμία αναφορά στην πρόταση του μοντέλου τη Νέα Ζηλανδία, στην οποία η κυβέρνηση συνεργάζεται με του παραγού και του διανομή για να ενθαρρύνει την παραγωγή ασφαλέστερων και δεόντω ελεγχόμενων λύσεων. Και δεν υπάρχει καμία σοβαρή αξιολόγηση των ωφελιών αυτού του μοντέλου για την προσαρμογή του στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν και είναι νωρί για να εκτιμηθεί συνολικά η αποτελεσματικότητα του μοντέλου τη Νέα Ζηλανδία, θεωρούμε ότι μια επανεξέταση των πολιτικών επιλογών για την αντιμετώπιση του πολύπλοκου φαινομένου των νέων ψυχοτρόπων ουσιών πρέπει να, να περιλαμβάνει μια σαφή αξιολόγηση βιωσιμότητα μια τέτοια προσέγγιση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από όσο γνωρίζω, η Επιτροπή έχει ήδη ενημερωθεί για ένα αντίστοιχο μοντέλο ρύθμιση παραγωγή και διάθεση κάναβη, τι λεγόμενε κοινωνικέ λέσει κάναβη και έχει δείξει ενδιαφέρον. Τα εμπειρικά στοιχεία μας δείχνουν ότι υπάρχουν πιθανές αναλλακτικές προτάσεις σε σχέση με την ποινικοποίηση που μπορούν να έχουν επιθυμητά αποτελέσματα για τις κοινωνίες και τις κυβερνήσεις, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αρνητικές συνέπειες ποινικοποίηση μεμονωμένων χρηστών. Ενώ οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες θέτουν νέες προκλήσεις για τα εφιστάμενα μοντέλα, μοντέλα ελέγχου των ναρκωτικών, η εμφάνισή τους παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να εξετάσουμε τη συνολική και επιλωτική δοκιμή εναλλακτικών μοντέλων πολιτικής και νομοθετικών προσεγγίσεων για τον έλεγχο των ναρκωτικών. Είναι απαραίτητη μια αντικειμενική εκτίμηση κόστου-οφέλου που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα για να αξιολογηθεί η χρησιμότητα των διαφορετικών μοντέλων ελέγχου καθώ και επιπτώσει στη δημόσια υγεία. Κεντρικό στόχο πρέπει να είναι η προστασία τη δημόσια υγεία και τη ευημερία των πολιτών. Σίγουρα η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά και συνεργασία μεταξύ, η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποφυγή Ασθενειών και Ελέγχου. Οι νέε ψυχοδραστικέ ουσίε δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν υπό το πρίσμα μια παρανομία, αλλά με διαφανεί νόμιμε ρυθμίσει και έλεγχο που θα του αφαιρέσουν τη γοητεία του απαγορευμένου και θα μειώσουν τη βλάβη στην κοινωνία του χρήση και την οικονομία. Ευχαριστούμε. Η Κομισιόν για να κλείσουμε. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Αντωνέσκου για, την ε, πολύ ε, για το πολύ επικοδομητικό σχέδιο γνωμοδότησης για τις νέε ψυχότροπες ουσίες. Ε, καλωσορίζουμε το γεγονό ότι η συγκέντρια συμμερίζεται τις ανησυχίε μα σε σχέση με τι προκλήσει που ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τι νέε αυτέ ουσίε. Χαιρόμαστε που επίση συμμερίζεται τι ανησυχίε για το ότι η ε, άμεση διάδοση αυτών των ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ιστορική τη αγορά αποτελεί πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί είναι, αποτελεί ευρωπαϊκή πρόκληση και πολύ γρήγορα να μιλήσω για τα αριθμητικά στοιχεία που μου αναφέρει. Όντω υπάρχουν όλο και περισσότερε ε, ψυχότροπε ουσίε στην Ευρώπη. Μιλούμε για 73 κοινοποιημένε από τα κράτη-μέλη πέρσι. Θα υπάρξουν τουλάχιστον ε, άλλε τόσε φέτο και συνολικά έχουμε περίπου 300 νέε ψυχότροπε ουσίε οι οποίε έχουν ε, αναδυθεί και πολλέ από αυτέ κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά. Που σημαίνει ότι υπάρχουν όλο και περισσότερε νέε ψυχότροπε ουσίε στην αγορά από ότι υπάρχουν παράνομα ναρκωτικά. Γιατί υπάρχουν μόνο 234 ε, ναρκωτικά τα οποία ε, τα διέπονται από τι διάφορε συμβάσει. Οπότε αντιμετωπίζουμε σημαντικό ε, πρόβλημα γιατί οι ψυχότροπες ουσίες αυξάνονται συνεχώ και είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα γιατί η ιστορική αγορά επιτρέπει σε αυτές τις, ε, ουσίες να κυκλοφορούν ελεύθερα και όντω κυκλοφορούν ελεύθερα. Όπω λέει και η συγκήτρια, 80% αυτών των ουσιών ε, υπάρχουν σε πάνω από ένα κράτος μέλος. Δεύτερον, καλωσορίζουμε το γεγονός ότι η συγκήτρια συμμερίζεται την άποψή μας ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ανταπόκριση στις προκλήσεις που, που θέτουν αυτές οι νέες ψυχότροπες ουσίες, γιατί αυτός είναι ακριβώς ο στόχος του προτινόμενου κανονισμού. Προετοιμα... Θέλουμε να ενισχύσουμε την ανταπόκριση μέσω ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, μέσω τη αξιολόγηση κινδύνου των ουσιών και μέσω ε, μιας μεγάλης πανοπλίας μέτρων που θα εισηχθούν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αυτός ο κανονισμός, ο προτινόμενο κανονισμός, έχει ως στόχο να παράσχει μια πιο αποτελεσματική και έξυπνη απάντηση στις προκλήσεις αυτών των ουσιών, διευκολύνοντας την ανάληψη δράσης πιο γρήγορα και σε πιο πρωτογενείς ε, φάσεις ε, της ε, παραγωγής αυτών των ουσιών, καθώς επίσης και την πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση ανάλογα με τον κίνδυνο που υπάρχει από αυτές τις ουσίες. Σύντομα λοιπόν, κλείνοντας να πω ότι καλωσορίζουμε το γεγονός ότι η έκθεση της κυρίας Αντωνέσκου είναι πολύ υποκοδομητική, πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον, προσπαθεί με πολύ επικοδομητικό τρόπο να ενισχύσει την πτυχή της δημόσιας υγείας, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί και τη, και λογική και το σκεπτικό της ε, πρότασης όπως έχει παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι η συγκήτρια, οι σκιώδες και η Επιτροπή σας θα παίξουν σημαντικό, χρήσιμο ρόλο για την ενίσχυση αυτής της πρότασης και για, την, ε, για να τονιστεί η πτυχή των, ε, της δημόσιας υγείας της πρότασης. Και βεβαίως συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή ότι η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα σημαντική για να αντιμετωπιστούν ε, οι προκλήσεις των νέων ψυχοτρόπων ουσιών, αλλά επιπλέον και ως ε, ε, συνοδευτικό μέτρο στην νομοθεσία πρέπει να επενδύσουμε σε προληπτικά μέτρα στην θεραπεία, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τους κινδύνους που υπάρχουν από αυτές τις ουσίες. Και βεβαίως έχουμε δεσμευθεί να δούμε και σε όλο τον κόσμο που βρίσκονται οι καλύτερες, οι βέλτιστες πρακτικές για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό το οποίο ακόμα εξελίσσεται και είναι καινούριο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο. Ο εκπρόσωπος της ε, εισηγήτριας ε, αποχωρεί, οπότε περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερής διάταξης. Und wir sind am Ende Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Σημείο 13. Μπόγκουσλαβ Σόνικ. Η συγητής παίρνει και αμέσως το λόγο. Dziękuję panie przewodniczący. Jest to opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μιλούμε για μια γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας για την αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων και των ποινών που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών όσον αφορά τον ορισμό των ναρκωτικών. Αυτό είναι ο επίσημος τίτλος αυτής της νομικής πράξης. Το θέμα της αντιμετώπισης των νέων ψυχοτρόπων ουσιών είναι βεβαίως μια τεράστια πρόκληση και αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά και την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Αυτές οι νέες ψυχοτρόπες ουσίες παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά ως παράνομες ουσίες και κυκλοφορούν και τίθενται σε εμπορία. Βεβαίως αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την δημοσία υγεία των πολιτών, κυρίως για τους νέους που αποτελούν την πλειοψηφία των χρηστών. Εμεί τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερες ζημιές στην ανθρώπινη υγεία, καθώς επίσης και περιπτώσει θανάτων που προέρχονται από την λήψη τέτοιων ή τη χρήση τέτοιων ουσιών. Και λόγω και του κινδύνου που υπάρχει στο εμπόριο αυτών των ουσιών και λόγω των όσων συμβαίνουν εκεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο ένα νέο νομικό πλαίσιο, γιατί η αγορά είναι πολύ ευέλικτη. Μόλις κάτι απαγορευτεί, η αγορά πάντα είναι σε θέση εκείνη τη στιγμή να δημιουργήσει, να βρει μια νέα ουσία η οποία θα αντικαταστήσει την απαγορευμένη, με μια διαφορετική χημική σύνθεση. Ε, νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για αυτά τα χαρακτηριστικά των για την αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων κτλ. Ε, είναι πολύ ε, σωστή. Μιλούμε για την ε, δημιουργία νέων φορέων που θα παρακολουθούν τις ουσίες αυτές, τους κινδύνους που, όπου ελοχεύουν για την, για την υγεία των πολιτών και επίσης μιλούμε ε, για τη συμπλήρωση του ορισμού των ναρκωτικών με τις ε, ε, ουσίες. Ε, επίσης, έχω σας κάνω και εγώ μια πρόταση. Ο ορισμός θα πρέπει να μιλά και για μείγματα ε, ουσιών πέραν των όσων περιλαμβάνει, σε, διάφορα, σε διάφορους συνδυασμούς γιατί οι ε, συνέπειε ε, των, ε, των ουσιών αυτών μπορούν να είναι πολύ διαφορετικές ανάλογα και με τη χημική του σύσταση. Νομίζω λοιπόν ότι τα μείγματα είναι πολύ σημαντική τροπολογία και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο, στο πρώτο εγώ λοιπόν. Και η πρόταση για τη διεύρυνση αυτού του, αυτής της απόφασης πλαισίου με αυτά τα με τα δικήματα τα λοιπά και τις ποινές. Νομίζω ότι πρέπει να τύχει ε, της υποστήριξής σας γιατί αυτές οι ουσίες είναι ιδιαίτερα ε, επικίνδυνες για την δημοσιογεία και πρέπει βεβαίως να ε, περιληφθούν και στον ποινικό κώδικα. Μέχρι τις 7 του Γενάρη μέχρι τις 5 το απόγευμα μπορείτε να στείλετε τις προτάσεις για τροπολογίες. Ο κύριος Χρυσόγελος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε συνέχεια και της προηγούμενης συζήτησης ε, νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών όπως εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια αν κρίνουμε από τα αποτελέσματά του έχει αποτύχει γιατί δεν έχει καταφέρει να μειώσει ούτε τη ζήτηση ούτε την προσφορά των παράνομων ουσιών ενώ έχει παράλληλα οδηγήσει σε αύξηση των βλαβών για την κοινωνία Όπω μα ενημερώνει και η έκθεση Reuter Trautmann που υλοποιήθηκε για λογαριασμό τη Επιτροπής το 2009. Χαρακτηριστικό αυτή τη αποτυχία είναι η συνεχώ αυξανόμενη εμφάνιση νέων επικίνδυνων συνθετικών και ε, φυτικών ψυχοδραστικών ουσιών που δεν υπάρχουν σε κανένα καθεστώ ελέγχου και συζητήσαμε μόλι πριν. Οι κατασταλτικέ πολιτικέ που εφαρμόζονται και η ποινικοποίηση των χρηστών έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά από τι ε, μεγαλύτερε ψήδιε ουσίε, όπω καταδεικνύουν πρόσφατε διεθνεί έρευνε που εξετάζουν το κόστο τη ποινικοποίηση των ουσιών και των χρηστών. Σύμφωνα με τι εκθέσει, ο πόλεμο κατά των ναρκωτικών και η ποινικοποίηση τη χρήση ουσιών, όπω εφαρμόζεται, απειλεί τη δημόσια υγεία, εξαπλώνει ασθένειε και προκαλεί χιλιάδε θανάτου, υποδαβλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, προωθεί τον κοινωνικό στιγματισμό και αποκλεισμό και ενισχύει την εγκληματικότητα, ενώ σπαταλάει δισεκατομμύρια σε μια αναποτελεσματική εφαρμογή του νόμου. Οι χρήστε των ουσιών, ιδιαίτερα οι προβληματικοί και αισθηματικοί, παρουσιάζουν σταθερέ τάσει, αλλά είναι πιο πολύ από ποτέ η προσφορά παραγωγή ουσιών έχει σταθερά αυξητικέ τάσει, καθώ και τα κέρδη από το οργανωμένο έγκλημα ή για το οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά, ενώ παρουσιάζονται ανησυχητικέ τάσει πολυτοξικομανία και διάδοση του ιού HIV ανάμεσα στου χρήστε ενδοφλέβιων ουσιών. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται το 2011 είχαν περισσότερο από 300 εκατομμύρια χρήστες παράνομων ουσιών, με αύξηση περίπου 18% μέσα στο 2008. Γεγονός που καθιστά αδιανόητη την αντίληψη να τους θεωρούμε όλους εγκληματίες. Οι κατασχεθήσεις ποσών του ουσιών είναι πιο πολλές από ποτέ, αλλά αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσό των παραγόμενων ποσοτήτων ουσιών. Από τι κυβερνήσει δαπανούνται υπέρογκα ποσάδες εκατομμυρίων σε μια αναποτελεσματική πολιτική αστυνόμευση και ελέγχου, το 80% των συνολικών δαπανών στοχεύει στην αστυνόμευση, ενώ μόνο το 20% στη θεραπεία και πρόληψη. Τα κέρδη όμως από το παράνομο εμπόριο έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, δηλαδή έχουν ξεπεράσει τα 400 δισεκατομμύρια σε αιτήσια βάση. Στη χώρα μου την Ελλάδα έχουμε μια δραματική αύξηση των κρουσμάτων διάδοσης του ιού HIV, ενώ απόρρια της φτώχειας, ενεργείας και των απογορευτικών πολιτικών έχουν εμφανιστεί νέε πολύ επικίνδυνες, αλλά φτηνές συνθετικέ ουσίε, όπως η ΣΥΣΑ που έχει στην κυριολεξία θερήσει τις πιάτσες των τοξικαμανών με καταστροφικές συνέπειες για την υγεία τους. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για τα Ναρκωτικά, η αγορά ναρκωτικών σήμερα δείχνει να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία και δυναμισμό και να στηρίζεται λιγότερο σε φυτική προέλευση ουσία. Τονίζεται ότι υπάρχει σημαντική αύξηση νέων συνθετικών ψυχοδραστικών ουσιών που δεν υπάγονται στο καθεστώ ελέγχου με δεδομένο ότι ένα στου τέσσερι Ευρωπαίου πολίτε, τουλάχιστον 85 εκατομμύρια άνθρωποι, έχει κάνει ή εξακολουθεί να κάνει χρήση παράνομων ουσιών, πρέπει να βρούμε πιο ανθρώπινου δίκαιου και αποτελεσματικού τρόπου για να αντιμετωπίσουμε τη χρήση και την εξάρτηση από ουσίε. Οι ασθένειε, η θάνατη και η κλιματικότητα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά θα αυξάνονται όσο αφήνουμε τι ουσίε χωρί έλεγχο και νόμιμη ρύθμιση στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματο. 80 χρόνια μετά τη λήξη από το απαγόρευση στην Αμερική αλλά και 50 χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου κατά των ναρκωτικών θα, θα, έχουμε, θα έπρεπε να έχουμε μάθει το μάθημά μας ότι μέσα από την απαγόρευση δεν μπορείς να ελέγξεις ούτε την προσφορά ούτε τη ζήτηση ουσιών και δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο μέσα από ένα καθεστώ παρανομία, δεν προστατεύει τους χρήστε, την υγεία και τα δικαιώματά του, ενώ η μαφία θησαυρίζει. Ένα από τα πιο σοβαρά και ανησυχητικά φαινόμενα απόρρια των πολιτικών αυτών είναι η πολιτικοκομανία που επικρατεί ιδιαίτερα ανάμεσα στην νεολαία, αλλά και η πρόθεση στην αγορά όλο και πιο επικίνδυνων νέων σιών που δεν, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν με απαγορεύσει που θα τι οδηγήσουν περαιτέρω υπόγεια στην παρανομία, αλλά με έμφαση στον έλεγχο, την νόμιμη ρύθμιση, τη μείωση τη βλάβη και τη προστασία τη υγεία και των θεμελιωδών δικαιωμάτων καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπερψηφίσει από το 2004 την έκθεση Κατάνια που όμως δεν έχει βρει το δρόμο της εφαρμογής ως ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική και είναι καιρός να ξαναδούμε σοβαρά τις συστάσεις αυτές. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει μια σοβαρή κινητικότητα από επιστήμονε, πολιτικού, ανθρώπου των τεχνών και των γραμμάτων για να υπάρξει αλλαγή των πολιτικών με έμφαση στη διασφάλιση δημόσια υγεία, των δικαιωμάτων των καταναλωτών ουσιών καθώ και των προγραμμάτων μείωση βλάβη, σταδιακή απεξάρτηση και επανένταξη στην κοινωνία στηριζόμενα στα επιστημονικά δεδομένα, την αντικειμενική πληροφόρηση και τι διεθνεί καλέ πρακτικέ, αντί για ιδεοληψίες και πολιτικέ πανικού. Ήδη στα Ηνωμένα Έθνη έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό ρεύμα από χώρε που επιστούν μια άλλη νόμιμη ρύθμιση παραγωγή και διάθεση ουσιών, με την Ουρογουάη να έγινε πρόσφατα η πρώτη χώρα παγκοσμίω που νομοποιεί την παραγωγή και διάθεση κάναβη με στόχο να περιορίσει το οργανωμένο έγκλημα και να προστατεύσει του καταναλωτέ στη χώρα τη. Πολλές πολιτείες στις ΗΠΑ ε, Πολιτείες Αμερικής έχουν ακολουθήσει παρόμοια τακτική και άλλες συνέτοιμες να ακολουθήσουν, ενώ και στην Ευρώπη όπου έχουν εφαρμοστεί εναλλακτικά μοντέλα ελέγχου και ρύθμιση των ουσιών, δηλαδή Πορτογαλία, Ελβετία, Ολλανδία, τα αποτελέσματα είναι σημαντικά και εντυπωσιακά. Χρειαζόμαστε λοιπόν άμεσα μια ρεαλιστική και αντικειμενική εκτίμηση του κόστου και τη αποτελεσματικότητα των κατασταλτικών πολιτικών που ακολουθούνται, αλλά και να εξετάσουμε σοβαρά εναλλακτικού τρόπου ρύθμιση και ελέγχου των ουσιών με βάση την επικινδυνότητά τους, το διαχωρισμό ε, της εμπορίας από τη χρήση, με έμφαση στη μείωση της βλάβης και την ε, αποποινικοποίηση της χρήσης ορισμένων. Ευχαριστούμε. Jut. ik moet eh, het voorstel nog eh, goed bestuderen. Ε, θα πρέπει να το δούμε, να, δω το θέμα με περισσότερες λεπτομέρειες και να το συζητήσω με την ομάδα μου. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα της νομοποίησης και της ποινικοποίησης. Ευχαριστώ. Uh, thank uh, Μιλώ εκ μέρους του συνάδελφου του Αντώνη που δεν κατάφερε να έρθει σήμερα. Ε, η κυρία Παρβάνοβα θέλει να ευχαριστήσει ε, τον ε, συγητή. Στόχος μας είναι η προστασία της δημοσίας υγείας. Ε, είναι πολύ θετική η οδηγία πλαίσιο του Συμβουλίου και η πρόταση περίθμησης των νέων ψυχοτρόπων Η... Το παρόν πλαίσιο, το ισχύον πλαίσιο, χρειάζεται ενημέρωση ίδια, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την, τον ορισμό του ναρκωτικού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες στη δημόσια υγεία. Ε, ομάδες και οργανωμένων κλίματος ε, έχουν τεράστια κέρδη από διακίνηση ναρκωτικών. Η αγορά ανέρχεται στα 70 δισεκατομμύρια σύμφωνα με εκτιμήσεις, ετησίως. Αυτά είναι έσοδα των παρανόμων οργανώσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει μέτρα εναντίον τη παραγωγή και διακίνηση. Δεδομένων των κερδών λοιπόν των αυτών των οργανώσεων ε, χρειάζεται να είμαστε πολύ πιο δραστήριοι. Είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε νομοθεσία αλλά και ε, αυτή η νομοθεσία να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία. και Παρβάνοβα θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον εισηγητή η διάταση ότι αφορά ε, τα θέματα απειλών ανησυχίας και τη δημόσια υγεία γενικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Κομισιόν για να κλείσουμε, αν θέλετε. Σύντομα. Many thanks, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας ε, τον εισηγητή, τον κύριο Σόνικ, για ένα πολύ επικοδομητικό σχέδιο έκθεσης ε, για την ε, οδηγία που τροποποιεί την οδηγία για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Το θέμα είναι η περισσότερο επιβλαβής να αντιμετωπίζονται ως στο πλαίσιο του, ε, των ποινικών πράξεων ε, ε, μιλάμε βέβαια και για τα ναρκωτικά, τα οποία βέβαια θα είναι θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ποινικών, του ποινικού δικαίου και αυτό γιατί είναι αποτρεπτικός ο χαρακτήρας του ποινικού δικαίου και πιστεύουμε ότι οι προτάσεις που έγιναν από τον κύριο Σόνικ σε σχέση με την ανάγκη διευκρίνησης ορισμένων διατάξεων της προτινόμενης οδηγίας και συγκεκριμένα να δοθεί περισσότερη έμβαση στα μείγματα ε, τέτοιων ε, νέων ουσιών. Είναι πιο επικοδομητικά τα σχόλια αυτά και πάρα πολύ ε, χρήσιμες οι προτάσεις αυτές. Εμείς ευχαριστούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να ενισχύσουμε την πρότασή μας αυτή. Ευχαριστούμε. Συγητής. E, να ευχαριστήσω την Κομισιόν να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους. Η ποινική δίωξη ε, που ανέφερε ο Έλληνας συνάδελφος, ε, πρέπει να πω ότι για τέσσερα χρόνια είχαμε ε, συζητήσει το θέμα αυτό για αυτά στις ψυχότροπες ουσίες που χρησιμοποιούνται κυρίως από νέους Γι' αυτό αποφασίσαμε το συντομότερο δυνατό να προχωρήσουμε τη δουλειά πάνω σε αυτή την οδηγία και θέλαμε κυρίως τα, τα μείγματα, τις μικτές ουσίες να τις καλύψουμε με τούτο τον κανονισμό, με τούτη τη διάταξη. Προθεσμία και τροπολογίε, όπως είπε ο συγητή, 7 Ιανουαρίου, 15, 17 το απόγευμα, 5 το απόγευμα. 30 Ιανουαρίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσουμε. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημέρας της διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων για την κλωνοποίηση. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο και ένα ψήφισμα ως προς αυτό. Η κυρία Ροθπέραντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι αντίθετη με την κλωνοποίηση. Οπότε θα πρέπει να, να φύγω και αμέσως στις 5.30 για να πάω στους, ε, στους συντονιστές και γι' αυτό θα πρέπει να κλωνοποιηθώ, αλλά που είμαι αντίθετη. Λοιπόν, υπάρχει ένα ψήφισμα εδώ διαφόρων ε, ε, συναδέλφων. Ουσιαστικά μιλούμε για αυτή την παλιά ιστορία Θυμόμαστε όλοι ε, αυτές τις ατυχείς ε, ε, συζητήσεις που κατέρευσαν γιατί η Κομισιόν δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε δήλωση για τον κλωνοποίηση και είχε υποσχεθεί, είχε πει τέλο πάντων ότι κάποια στιγμή θα έρθει με μια νομοθετική πρόταση. Ακόμα περιμένουμε αυτή την νομοθετική πρόταση και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την επισήμανση του βοηού κρέατος είπαμε πολλές φορές ότι θέλουμε να υπάρχει μια δήλωση, μια αναφορά για το πότε τέλος πάντων θα έρθει αυτή η νομοθετική ε, πρόταση. Ε, υπάρχει γι' αυτό λοιπόν η ε, προφορική ερώτηση που θέτουμε. Μέχρι στιγμής απάντηση δεν έχουμε πάρει. Υπάρχουν διάφορες φήμες που κυκλοφορούν, που υπήρχαν και από τότε με την επισήμανση του βοήου. Τότε υπήρχαν σαφείς δηλώσεις, εδώ και ένα μισό χρόνο δηλαδή, που κατέρευσαν οι συζητήσεις ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας το, στην ιστοσελίδα του δημοσίευσε ότι ε, ε, δεν χρειάζεται κανένας να ανησυχεί στις ΕΙΠΑ γιατί θα απαγορευτεί η κλωνοποίηση ε, αλλά καμία τέτοια πρόταση δεν είδαμε αντιστοίχως από την Κομισιόν. Ε, κάναμε λοιπόν ε, αυτό το ερώτημα προς την Κομισιόν, να μας πει η Κομισιόν τι προτίθεται να κάνει, Κομισιόν πείτε μας τι θέλετε να υποβάλλετε ως πρόταση, τι κάνατε στο παρελθόν, κάνατε αξιολόγηση επιπτώσεων, γιατί δεν τη δημοσιεύσατε, η θέση σας ποια είναι τώρα για την ε, υποχρεωτική επισήμανση, ε, κυρίως για τα, ε, για τα ζώα που έχουν γεννήσει κλωνοποιημένα. Ε, όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Γιατί ο ε, Επίτροπος Εμπορίου, ο Ντεχούχτ, έχει διαφορετική άποψη ε, ίσως από, τους, ε, από τον Επιτροπό για τους καταναλωτές. Αυτό δεν θα μας εξέβλητε. Επίσης, θέλουμε να μάθουμε από την Κομισιόν, αν θέλει να δεσμευθεί, ε, να κάνει μια δήλωση για τις διαπραγματεύσεις της εμπορικές. Τώρα, έχουμε ακούσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, αν όχι τούτη τη βδομάδα, την επόμενη βδομάδα θα υποβάλει κάτι. Ε, κοιτάω προς την Κομισιόν, βλέπω τους ε, κυρίως από την Κομισιόν, τους εκπροσώπους. Αν όντω λοιπόν υποβάλλει κάτι την επόμενη εβδομάδα η Κομισιόν, ε, δύο πράγματα θέλω να πω εγώ. Ε, ρωτάμε εδώ και πολύ καιρό. Δεν θα ήταν πιο ευγενικό έτσι, αυτό το παλιωμοδίτικο, αυτή της παλιωμοδίτικης ε, ευγένεια να μας δείγμα, να μας ε, ενημέρωνε η Κομισιόν για το τι κάνει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αποφασίσει κάτι η Κομισιόν πριν τα α, Χριστούγεννα, αλλά αν όντω κάνει κάτι, έχω μια πρόταση εδώ στα χέρια μου και στην πρόταση λέει διάφορα πράγματα τα οποία όμως δεν βρίσκω καθόλου ενδιαφέροντα. Στην πρόταση της Κομισιόν υπάρχουν δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Μία πρόταση για οδηγία, για την κλωνοποίηση των ε, ε, ζώων, ε, των βοηδών και μία πρόταση για την θέση σε εμπορία. Αλλά τίποτα ουσιώδες δεν υπάρχει. Στο άρθρο 3 λέει τι απαγορεύεται στα κράτη-μέλη. Η κλωνοποίηση των ζώων, και η θέση σε εμπορία κλωνοποιημένων ζώων και των εμβρίων. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο που να έχει να κάνει με τις επόμενες γενιές. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Γενικώ τίποτα. Πάμε τώρα στο κομμάτι της θέσης εμπορία τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Η Κομισιόν τι έπρεπε να προτείνει ως προς αυτό, ε, που δεν το έκανε γιατί θα έπρεπε να μας έχει ενημερώσει. Εκεί λοιπόν στο άρθρο 3 πάλι λέει ε, απαγορεύσεις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα δεν τίθεται σε εμπορία. Τελεία. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το, τα τρόφιμα ε, ζωικής προέλευσης που εισάγονται από τρίτες χώρες όπου μπορεί να υπάρχει νόμιμη θέση εμπορία ε, κλωνοποιημένων ζώων τίθονται σε εμπορία, τίθονται σε εμπορία στην Ένωση μόνο σύμφωνα με συγκεκριμένε διατάξεις ε, εισαγωγών που αναφέρονται στον, αρθρο 48 48-49 του κανονισμού ΤΑΔΕ. Τι σημαίνει αυτό κύριε Πρόεδρε? Όποιο βρίσκεται στην ε, Αμερική, στην Κίνα που θέλει νομίμως να ε, κλωνοποιήσει μπορεί ωραιότατα να στείλει τα, ε, το κρέα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον δεν χρειάζεται καμία επισήμανση. Ειλικρινά. Ε, λυπούμε. Ε, Ήθελα να ξεκινήσω τις διακοπές μου με ηρεμία, αλλά δεν θα τα καταφέρω. Αν όντως ε, υπάρχει κάτι αληθινό σε αυτά που υπάρχουν στην πρόταση, πραγματικά μιλάμε για σκάνδαλο και η Κομισιόν δεν καταλαβαίνει. Αν θέλετε να κάνετε δώρα στους, ε, στους Αμερικανούς, κάντε τους πιο έξυπνο δώρο. Το, είναι καλό το σύστημα, το, το χρονικό σημείο. Ε, δε, ελπίζετε, ίσως ε, αδίκως ότι το νέο κοινοβούλιο δεν μπορεί να μην ξέρει τι ακριβώς να κάνει με την πρόταση αυτή. πρέπει να σας πω ότι πολλοί από τους ε, συναδέλφους, ε, εγώ δεν θα είμαι εδώ, αλλά πολλοί από τους συναδέλφους που θα είναι εδώ ε, θα το παρακολουθούν το θέμα αυτό, γιατί πραγματικά είναι εσχρό αυτό που γίνεται. δεν θέλουμε κλωνοποίηση των ζώων. Δεν θέλουμε να μπαίνουν σε θέσεις εμπορία για την παραγωγή τροφίμων. Και αυτό το, το νέο, αυτή η είδηση δεν έχει φτάσει στην Κομισιόν. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Πραγματικά, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο. Εγώ θέλω να στείλουμε ένα ξεκάθαρο α, μήνυμα. Η Κομισιόν πραγματικά ε, είναι εσχρό αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή και δεν θα πρέπει να το συνεχίσει. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Έχουμε απόφαση των συντονιστών ότι θα στείλουμε μία επιστολή. Την κάναμε, τη στείλαμε. Και Ελπίζουμε ότι η πρόταση Κομισιόν δεν θα, είναι, θα έρθει μετά από όλα όσα έγιναν ε, ε, μετά από εκείνες τις ε, διαπραγματεύσεις που κατέρευσαν. Όπως είπε λοιπόν και η Ντάγμαρ, πραγματικά είναι κάζους μπέλι αυτό για το Κοινοβούλιο. Προχωρούμε στη συζήτηση. Κύριε Λεπάζ. Stevenson und Peter Κύριε Πρόεδρε, δεν θα σας κάνει εντύπωση ότι συμμερίζομαι την αγανάκτηση την οποία μόλις εξέφρασε η κυρία Ροτ Μπέρεντ. Τα δύο έγγραφα τα οποία έλαβα πριν από 10 λεπτά είναι απαράδεκτα, είναι αδύνατο να τα δεχθεί κανείς δεν μπορώ να περιγράψω τι αισθάνομαι. Πριν από μερικά χρόνια το Κοινοβούλιο ψήφισε ότι δεν θέλει κλωνοποίηση. Το είχαμε πει σαφέστατα. Είχαμε συζητήσεις, δείξαμε καλή θέληση, ε, θα το θυμάστε, προσπαθήσαμε να βρούμε μία λύση ε, συνενετική το κείμενο που λάβαμε σήμερα το απόγευμα δεν προβλέπει καθόλου την ενημέρωση του καταναλωτή. Είναι πολύ απλή ερώτησή μου κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε οριστικά η παραγωγή της κτηνοτροφίας ε, να σημαίνει δυσπιστία ε, από πλευράς καταναλωτή με όλες τις, ε, τα σκάνδαλα που ζήσαμε τα διατροφικά για να δώσει τη δυνατότητα στο βραζιλιάνικο, αργεντίνικο, αμερικανικό κρέας ε, να αντικαταστήσει το ευρωπαϊκό κρέας ή είναι σοβαρή. Και αν είναι σοβαρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι δυνατόν να μας προτείνει ένα τέτοιο είδους κείμενο, το οποίο είναι απαράδεκτο για του συμπολίτε μας ήδη η τεράστια πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν θέλει να καταναλώνει ε, κρέας ε, κλωνοποιημένο ή από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας δεν τον θέλουν. Αν δεν τους δίνετε τη δυνατότητα μέσω της αγοράς με την κατάλληλη ετικετοθεσία να, γνωρίζουν τι ακριβώς καταναλώνουν, είναι πολύ απλό αυτό. Δεν πρόκειται να καταναλώσουν πλέον και θα έχουμε μια νέα κρίση κτηνοτροφική στην Ευρώπη που θα είναι βέβαια ε, ίδια με αυτήν που έχουμε ζήσει στο παρελθόν και μου κάνει εντύπωση, θα μου κάνει εντύπωση να έχει τέτοιου είδους στόχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λεπάζ. Ο κύριος Στάς δεν είναι εδώ. Η κυρία Λιωτάρ. Ως ε, Εισηγήτρια και εγώ θα καταλαβαίνετε ότι παρακολουθώ το θέμα της κλωνοποίησης ε, πολύ στενά. Από το Μάρτιο του 2011 με τον αποτυχημένο τριμερή διάλογο ε, όπως γνωρίζετε είμαι εναντίον της κλωνοποίησης των ζώων Η σε ό,τι αφορά το κρέας των ζώων. Η πλειοψηφία των καταναλωτών διαφωνεί με το να παίζουμε με τη φύση με αυτόν τον τρόπο. Το Κοινοβούλιο ήταν στο παρελθόν πολύ σαφές στα μηνύματά του. Πέραν του ηθικού ζητήματος ε, υπάρχει και το ζήτημα της υγείας. Ε, η Κομισιόν στον τριμμένο διάλογο για τα νέα τρόφιμα για τα οποία η συγκήτρια προσπάθησε να επιτύχει ένα συμβασμό αλλά δεν έγινε κατορθωτό. Ήταν μια προσπάθεια τελευταία στιγμής ε, ε, το Κοινοβούλιο ήθελε μια συμφωνία, αλλά δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε αποδυνάμωση του κειμένου, δεν θα έφερνε πουδενή κέρδη για τους καταναλωτές. Νομίζω ότι η Κομισιόν ε, μας έφερε μια πρόταση που πραγματικά υπολείπεται τις θέσεις του Κοινοβουλίου, δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε ε, το κείμενο αυτό που έφερε στον τριμερή διάλογο η Κομισιόν. Και προφανώς δεν υπάρχουν μυστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα δύο έγγραφα θα γίνουν και αυτά γνωστά, θα ε, δημοσιοποιηθούν και ελπίζω η Κομισιόν να διαψεύσει ότι είναι πρόταση που προτίθεται να υποβάλει. Είναι εκπληκτικό που αυτή είναι η πρόταση μετά από τόσο χρόνο που ε, περιμέναμε μια απαγόρευση στην ε, παραγωγή και την εμπορία κλωνοποιημένων προϊόντων. Αυτά τα ε, έγγραφα δεν μιλούν καθόλου για κατιόντα, δεν περιλαμβάνουν απαγόρευση. Προφανώς δεν είναι η επίσημη εκδοχή αλλά από ό,τι βλέπω η Κομισιόν το μόνο που σκέφτεται είναι ο, οι διατλαντικές εμπορικές ροές και τίποτα άλλο. Δεν μιλούμε καν για, για τις επόμενες γενιές, ε, δεν αναφέρεται τίποτα για τα κατιόντα ζώα. με ανησυχή η ποιότητα της ε, νομοθεσίας μας. Η Κομισιόν προφανώς αγνοεί τα πραγματικά προβλήματα, ε, αγνοεί το θέμα των ε, κατιόντων ζώων, δηλαδή των γόνων ζώων που έχουν κλωνοποιηθεί, η Κομισιόν απλώς εφαρμόζει κάποια νομοτεχνικά κόλπα χρησιμοποιεί το 352 αντί του 114 κάτι που σημαίνει ότι το κοινοβούλιο δεν μπορεί να υποβάλει τροπολογίες μπορεί μόνο να ε, συνεισφέρει με ένα ναι με ένα όχι η πρόταση αυτή λοιπόν είναι άχρηστη και αν η Κομισιόν πραγματικά θέλει να συνεργαστεί μαζί μας δεν είναι ο πιο σωστός ε, τρόπος και σίγουρα δεν είναι και καλύτερη προσέγγιση ό,τι αφορά τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Ο Στίβενσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θυμάμαι νύχτα να γίνεται εκείνος ο τριμερής διάλογος ε, για τα νέα συστατικά ε, τροφίμων πριν από τρία χρόνια και αυτό που κάναμε, που προσπαθούσαμε να κάνουμε, προσπαθήσαμε κάπως έτσι να δείξουμε ο καθένας τη δύναμή του και προφανώς όλη η δουλειά πήγε χαμένη γιατί καταλήξαμε στο να μην υπάρχει συμφωνία και δεν θα ήθελα να υπάρξει μια τέτοιου είδου κατάσταση ξανά. Ένας από τους, λίγου, από τους λόγους, παρά το γεγονός ότι συμφωνώ ε, με όλα αυτά που είπε η Ντάγμαρ ε, και οι άλλοι συνάδελφοι, νομίζω ότι ένας από τους λόγους ήταν ε, το μη πρακτικό της προτάσεως. Εμείς μιλούσαμε για μια απαγόρευση ε, απογόνων, ε, κρέατος απογόνων των των άμεσων απογόνων αλλά και μελλοντικών απογόνων των ε, αυτών και του κρέας που ε, προ, προκύπτει. Βέβαια, οι κτηνοτρόφοι λένε ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για κίνδυνο για την υγεία τουλάχιστον οι Βρετανοί λένε ότι ε, τα προϊόντα των ε, απογόνων των κλωνοποιημένων οργανισμών δεν δημιουργούν κίνδυνο για την θυμόσια υγεία. Δεν ξέρω λοιπόν, αν μπορούμε λοιπόν να εισαγάγουμε την ετικετοθεσία, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπορούμε να ζητάμε την απαγόρευση της κλωνοποίησης της χρήσης των, ε, του κρέατος των κλωνοποιημένων. Θυμάμαι τότε ότι ο πίτροπος είχε πει επειδή οι Αμερικάνοι δεν είχαν ανιχνευσιμότητα και ε, δεν είχαν και ποτέ, κατά τη γνώμη τους δεν υπάρχει κίνδυνος, αν εμείς επιβάλλουμε απαγόρευση θα σημαίνει έναν εμπορικό ε, πόλεμο που θα κάνει τον πόλεμο της μπανάνας πριν από 10 χρόνια να φαίνεται ε, κάτι το απολύτως ασήμαντο. Οπότε νομίζω ότι αν εμείς βάλουμε μία κόκκινη γραμμή και πούμε ότι τέτοιου είδους ε, ε, κρέας ε, δεν θα εισάγεται ή θα πούμε κάτι αντίστοιχο για τα προϊόντα που θα προκύπτουν από την Ευρώπη και δεν μπορούμε να τα εξάγουμε στις ΗΠΑ, νομίζω θα προκύψει ένας εμπορικός πόλεμος. Αν λέμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος για τους κατανάλωτες στην Ευρώπη όταν καταναλώνουν κρέας από κλωνοποιημένα ζώα, Χρειαζόμαστε επιστημονικά στοιχεία. Και αν οι Βρετανοί κτηνοτρόφοι αλλά και η Συνομοσπονδία Κτηνοτρόφων της Ευρώπης λένε ότι τα κλωνοποιημένα προϊόντα στη διατροφική αλυσίδα είναι ασφαλή, από πού προέρχονται αυτά τα επιστημονικά στοιχεία. Ας δούμε τα πράγματα πως έχουν. Καταλαβαίνω ότι οι συντονιστές έφτασαν ε, σε συμφωνία και καταλαβαίνω την ε, κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βασιστεί και σε επιστημονικά στοιχεία. Και εφόσον δεν έχουμε τέτοιου είδους στοιχεία και εφόσον δεν έχουμε κανένα άλλο πρακτικό τρόπο να επιτύχουμε την απαγόρευση που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να αφορά ε, την πρώτη γενεά ε, των κλωνοποιημένων ζώων, νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου θα καταλήξουμε τελικά σε κατάρρευση όλων των προσπαθειών μας. Γι' αυτό ελπίζω αυτή τη φορά να επιδείξουμε λίγο κοινή λογική, κύριε Πρόεδρε. Ο Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Ζόμερ που είναι υπεύθυνη για το ψήφισμα από την ομάδα μα. Ε, Δυστυχώ υπήρξε κάποιο ε, θάνατο στην οικογένεια, οπότε δεν μπορούσε να έρθει. Ε, εξ ονόματο λοιπόν τη κυρία Ζόμερ, αλλά και εκ μέρου μου, να πω το εξή. Έχω πληροφορίε ότι όντω η, πληροφορία, η έκθεση, συγγνώμη, η πρόταση θα έρθει την Τετάρτη. Μάλλον όμω δεν θα έρθει έτσι όπω ακούσαμε. φοβούμαι ότι η κατάσταση είναι άσχημη. Ελπίζω ότι δεν είναι τόσο άσχημη όσο νομίζουμε ή όσο περιμένουμε. Ε, από τις πληροφορίες μου, ο Επίτροπος Μπόργκ έχει προσπαθήσει πάρα πολύ να καταλήξει σε μια θέση που ε, θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο εκκίνησης της συζήτησης για το Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε να είναι λογική ως ε, βάση κίνηση, αλλά δυστυχώς η Κομισιόν δεν έδωσε την απαραίτητη στήριξη. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν αν σας αφορά η κριτική που ε, γίνεται θα πρέπει να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό γιατί ε, και εσείς ήσασταν ε, πρόσωπο της Κομισιόν, υπάλληλο της Κομισιόν όταν έγινε η πρόταση πριν από τρία χρόνια της Κομισιόν. Τότε που τη συζητούσαμε και την υποβάλατε μέσα στη νύχτα. Ούτως ή άλλως δεν είναι κακή. Ξέρω βεβαίως ότι υπήρξαν διάφοροι επίτροποι, διάφορες υπηρεσίες της Κομισιόν που ήταν ε, αντίθετη με την θέση του Κοινοβουλίου και ε, πρέπει να ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο το ξέρει αυτό. Ε, τώρα, για τη ΣΥΠΑ. Αν θέλουμε ελεύθερη συμφωνία εμπορίου με, το, με, το, με τη ΣΥΠΑ και καταλήγουμε σε τέτοια, σε τέτοια πρόταση, έμεινε μην απορρίτω όταν κάνουν εκστρατείες οι πολίτες στην Ευρώπη θέλουμε προστασία από το κλωνοποιημένο κρέας. Ε, προφανώς ε, θα αντιδράσει ο πολίτης. Πρέπει λοιπόν, ε, θα, προφανώς θα είναι αντίθετος με αυτή την ελεύθερη εμπορική, ε, με την ε, Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Πρέπει βεβαίως να συζητήσουμε μαζί με τους ε, πολίτες. Αλλά αν η Κομισιόν υποβάλλει κάτι τέτοιο μόνο και μόνο γιατί θέλει να καταλήξει με μια, σε μια Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τη ΣΥΠΑ, ε, μετά μπορείτε να καταλάβετε πώς θα είναι η συζήτηση και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Προσπαθήστε περισσότερο λοιπόν. Τώρα, για αυτό που είπε ο κύριος Στίβενσον. Σωστό, δεν υπάρχουν συγκεκριμένε επιστημονικέ αποδείξει ή στοιχεία ότι το ε, κρέα από κλωνοποιημένα ε, ζώα ή από την πρώτη γενιά ε, κλωνοποιημένου ζώου είναι βλαβερό. Αλλά βεβαίω η Κομισιόν λέει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερε μελέτε. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί είναι πολύ ε, θερμό θέμα. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι είμαι σίγουρος ότι δεν είναι βλαβερό. Όλοι λέμε μάλλον δεν είναι βλαβερό και μάλλον δεν υπάρχει λόγος πανικού. Αλλά υπάρχουν και θέματα υπέρ της προστασίας του, του, των ζώων, τα οποία συζητούνται και στον ε, ε, ΠΟΕ, συζητούνται και εδώ και πώς μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Δεν μπορούμε. Αν λοιπόν συμφωνούμε ότι ε, μιλούμε για την πρώτη ε, γενιά των ε, ζώων, θα πρέπει να δράσουμε δυναμικά. Στην διαδικασία συμφιλίωσης που έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο ήταν συγκεκριμένο το αίτημα. Αυτό τώρα που έχουμε, αυτό που ζητήσαμε μάλλον με την επιστολή των συντονιστών, ήταν πέραν του, της συναισθηματικής προσέγγισης του θέμα. Ήμασταν πολύ διπλωματικοί στην ε, διατύπωσή μας. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα χρειάζεται για την πρώτη γενιά των ζώων αυτών ε, μια συγκεκριμένη διάταξη. Και δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λέει η συνάδελφος, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε τροπολογίες. Εγώ τι θα πω στην, στην ομάδα μου. Υπάρχουν άλλες, άλλες εκθέσεις όπως η εκθεσού κουνή που σχετίζονται με αυτή την έκθεση. θα θυμώσουν και οι συνάδελφοι δηλαδή δεν μπορούμε κάθε, δυνατότητα, κάθε διαδικασία ε, να την αφήνουμε να καταραίει. Τότε λοιπόν μέσα στη νύχτα όταν συζητούσαμε δεν είχαμε δυστυχώς ε, τότε την ε, στήριξη της γερμανικής κυβέρνησης. Είχα έρθει εγώ πολλές φορές σε επαφή τηλεφωνική με την τότε Υπουργό Εμπορίου και μου είπε ότι εγώ προσωπικά είμαι υπέρ τη θέση του Κοινοβουλίου, αλλά υπήρξε, ήταν ε, ε ο Υπουργό Οικονομικών και δεν υπήρχε συμφωνία. Τώρα έχουμε μία νέα διατύπωση. Η ε, Γερμανία είναι υπέρ της απαγόρευσης ε, της κλωνοποίησης και της, είναι υπέρ της επισήμανσης των επόμενων γενεών. ελπίζω ότι θα βοηθήσει αυτό. Τότε δεν βοήθησε την Κομισιόν, ελπίζω τώρα να βοηθήσει και ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε και τροπολογίες στην διαδικασία της συναπόφασης. Αλλιώς ε, τα βλέπω πολύ μαύρα τα πράγματα και για τούτη την έκθεση και για άλλες και θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Αν θέλουμε ε, ε, συμφωνία ελεύθερου μπορείου με τους Αμερικανούς θα πρέπει καταρχάς να πάρουμε σοβαρά υπόψη μας το, τις ανησυχίες του, των πολιτών. Αν θέλουμε απλώς να καταστρέψουμε τα πάντα συνεχίζει η Κομισιόν να υποβάλλει τέτοιες προτάσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε άλλον έναν συνάδελφο, τον κύριο Χρυσόγελο. Πρέπει δυστυχώς να φύγω εγώ, ε, γιατί πρέπει να πάω στον ε, τριμερή διάλογο για το καπνό. Να πω ότι αυτή δεν είναι η πρώτη συμφωνία που καταλήγει σε κατάρρευση. Αν έρχονται τέτοιες προτάσεις ε, και συζητούμε τέτοια θέματα, πραγματικά θα πρέπει να βάλουμε ένα ένα ερωτηματικό, γιατί έχουμε εδώ ένα ε, κοινοβούλιο το οποίο <laughs> πραγματικά θα διασκεδάσει τους επόμενους μήνες με αυτές τις προτάσεις που έρχονται. Έχουμε ρωτήσει πολλές φορές πληροφορίες από την Κομισιόν πότε θα λάβουμε την ε, έκθεση. Πραγματικά είναι ένα κόλαφο στο, στο πρόσωπο των ε, καταναλωτών αν έρθει όντω τέτοια πρόταση έτσι όπως μας την παρουσιάζουν οι συνάδελφοι. Και νομίζω ότι αν θέλουμε ε, αποδοχή για το οικοδόμημα το ευρωπαϊκό, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες, ε, ε, τέτοιες προτάσεις, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που ερχόμαστε σε άμεση επαφή με, τους, με, τους, με αυτούς τους οποίους αφορά αυτή η πρόταση, με τους καταναλωτές δηλαδή. Πραγματικά πρέπει να το πάρουμε λοιπόν σοβαρά υπόψη μας και οι συνάδελφοι νομίζω ότι είναι έτοιμοι να δράσουν γιατί αλλιώς θα υπάρξει πραγματικά σοβαρό πρόβλημα μεταξύ Κομισιόν και, ε, και Κοινοβουλίου. Μιλώ ήραμα όπως βλέπετε, αλλά όντως θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Ο κύριος Γκρεμπράντη θα αναλάβει την Προεδρία και ο κύριος Χρυσόγελος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που στάμε, γιατί το θέμα των κλωνοποιημένων ζώων αφορά και τους καταναλωτές και τους κτηνοτρόφους και την οικονομία της Ευρώπης και την υγεία. Ε, ναι, σίγουρα θέλουμε εμπορικές σχέσεις, αλλά αυτές δεν είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή, οι εμπορικές σχέσεις πρέπει να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο που εξασφαλίζουν και το περιβάλλον και την υγεία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Επομένως, δεν θα προσαρμοστούμε ε, σε όρους ενός εμπορίου που δεν διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών Πιθανά θέλουμε τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και με άλλες χώρες, αλλά αυτές θα πρέπει να προσαρμοστούν στα υψηλά στάνταρτς τα οποία ζητάμε και για το περιβάλλον και για τους καταναλωτές και για την υγεία. Οποιασδήποτε επιλογές προωθεί η Κομισιόν, αν ισχύουν όσα είπαν πριν και οι συνάδελφοι, ε, δεν θα πρέπει να πλήξουν τους κτηνοτρόφους, το εμπόριο στην Ευρώπη, την υγεία των καταναλωτών και κυρίως την πίση των καταναλωτών ότι είναι ασφαλής καταναλώντας προϊόντα. Υπενθυμίζω ότι η αρχή που πρέπει να διέπει ε, τις αποφάσεις μας είναι η αρχή της πρόληψης. Δεν είναι η αρχή ότι νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις, νομίζουμε ότι ε, δεν πρέπει να περιμένουμε να αποδείξει κάποιος ότι τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από κλινοποίηση ή από απογόνους κλινοποιημένων ζώων είναι επικίνδυνα, αλλά είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει επίπτωση από την ε, κατανάλωση κλωνοποιημένων ζώων και απογόνων κλωνοποιημένων ζώων. Είναι διαφορετική η προσέγγιση, επομένως. Και επίσης βέβαια πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τα θέματα των δικαιωμάτων των ζώων και της προστασίας των ζώων. Νομίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο σωστά έχει διατυπώσει την άποψή του για απαγόρευση της κλωνοποίησης και της κατανάλωσης προϊόντων από κλωνοποίηση και από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων. Και το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει σήμανση εφόσον υπάρχουν προϊόντα τα οποία μπορεί να προέρχονται από κλινοποίηση ή από απογόνους κλινοποιημένων ζώων. Δεν μπορεί να είναι δικαιολογία ότι στην Αμερική δεν υπάρχει σύστημα ανείχνευσης, ανείχνευσιμότητας δηλαδή αν τα ζώα προέρχονται από κλόνους ή από απογόνους κλόνων. Δεν μπορεί σε αυτή τη βάση να αναπτύξουμε σχέση με τις ΗΠΑ. Και νομίζω ότι δεν πρέπει οι πολίτες και ενώπιση των ευρωεκλογών να σχηματίσουν την εντύπωση ότι αποδομούνται πολλά πράγματα στην Ευρώπη που βασίζονταν σε αξίες και σε αποφάσεις και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως είναι η προστασία από, τα, από, τους κλόνους και τους απογόνους κλόνων ζώων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χρυσόγελα. Μέχρι τώρα αυτό το... Τώρα ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό της ε, κλωνοποίησης των ζώων, αλλά βέβαια πρέπει να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από όλη την κριτική που άκουσε, κόντεψα να την ξεχάσω κιόλας. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε το λόγο για μια δύσκολη συζήτηση. Ακούσαμε όλες τις κριτικές, τις αυστηρές που απευθύνατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ο κύριος Λίζε συνόψισε το πώς αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει. Ξέρετε ότι υπήρξε μια πρώτη συζήτηση προσανατολισμού στις 27 Νοεμβρίου στο Σώμα των Επιτρόπων ε, και ε, το Σώμα θα αποφασίσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν ε, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο σε δύο μέρες, στις 18 Δεκεμβρίου δηλαδή. Δεν ξέρω ε, ποια είναι τα έγγραφα που λάβατε εσείς, ε, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα ήταν αντικείμενο ανεξέλεγκτης διαρροής, ε, γιατί είναι ακόμη εμπιστευτικά αυτά τα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, γιατί έγιναν συζητήσεις σήμερα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις 18 του μηνός θα αποφασίσουν οι επίτροποι, αλλά ίσως να έχετε και τα σωστά έγγραφα, δεν ξέρω, τα τα οποία τα λάβατε κάπως. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς την απόφαση των επιτρόπων σε δύο μέρες, αλλά είναι γεγονός ότι το έδειξε και η συζήτηση προσανατολισμού. Στο πλαίσιο της Επιτροπής υπήρχαν πολλές ε, φυγόκεντρες δυνάμεις ε, για διάφορους λόγους που φαντάζομαι τους καταλαβαίνετε. Θα καταλαβαίνετε επίση ότι είναι εμπιστευτικέ οι εσωτερικές συζητήσεις της ε, Επιτροπής, ε, του Σώματος των Επιτρόπων και εγώ δεν θα είμαι υπεύθυνο της διαρροή τους, αλλά θα ήθελα να πω στον κύριο Μπάνκι ότι το Νοέμβριο του 2012 ο Επίτροπος είχε έρθει και είχε υποσχεθεί να υποβάλει προτάσεις σε σχέση με ε, αυτά τα νέα συστατικά τροφίμων και την κλωνοποίηση των ζώων ε, ε, μέχρι τον ε, Ιούνιο του 2013, όμως έχουμε καθυστερήσει 6 μήνες, ελπίζω να γίνει αυτό, αν τα αποφασίσουν βέβαια οι Επίτροποι. Αυτοί οι 6 μήνες βέβαια δεν είναι λόγω λιγορίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά λόγω των ε, έντονων συζητήσεων που υπήρξαν στο πλαίσιο των εσωτερικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν μια πολύ δύσκολη συζήτηση Δεν θα σας τα αποκαλύψω όλα βέβαια, αλλά νομίζω ότι η ανάλυση του κυρίου Λίζε ήταν σχετικό ορθή. Υπήρξαν πολλές αποκλίσεις στο πλαίσιο των εσωτερικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, στο ψήφισμά σας μιλάτε για την ε, μελέτη επιπτώσεων που έγινε, θα δημοσιευθεί μαζί με τις προτάσεις Λίγες ημέρες μετά από την Τετάρτη τις λάβετε. Αλλά θα δείτε, υπάρχουν κάποια όρια. Δηλαδή, ο οικονομικός αντίκτυπος ως προς την πρακτική της κλωνοποίησης ε, στις ε, χώρες της Βορείου Αμερικής αλλά και της Νότιας Αμερικής είναι δύσκολο να αξιολογηθούν γιατί είναι ιδιωτικές δράσεις οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο ε, των δημοσίων αρχών της Αμερικής. Οι χώρες αυτές λοιπόν είναι πολύ διστακτικές, έχουν ενδιασμούς ως προς την αποκάλυψη οικονομική πληροφοριών σε σχέση με τον αριθμό των, ε, ε, των ε, κλώνων και του, της, του όγκου του κρέατος που προκύπτει από την κλωνοποίηση αυτή. Η συνδιαλλαγή του Μαρτίου του 2011 είχε αποτύχει όχι εξαιτίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά της απόκληση απόψεων, πιστεύουμε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με προτάσεις πολύ φιλόδοξες από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ πιο με, μετριασμένες από πλευράς Συμβουλίου και μεταξύ αυτών των δύο λοιπόν από απόψεων είχε αποτύχει στην διαλλαγή του Μαρτίου του 2011. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αρκετά ανοιχτή, ε, για μια πρόταση ενδιάμεση, κάπως μετριασμένη για να το πω έτσι. Ε, ο πρόεδρος Χρότε ξαναέγραψε στον ε, Επίτροπο. Ο Επίτροπος Μπόρζα έχει σκοπό από την Τετάρτη και μετά να του απαντήσει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το Σώμα των Επιτρόπων θα έχει αποφασίσει. Δεν θέλει να προκαταβάλει την ε, απόφαση των επιτρόπων, γιατί θα ήταν λίγο ε, γελίο να γίνει κάτι τέτοιο, να απαντήσει κανείς ε, στον ε, πρόεδρο της Επιτροπής σας, αν δεν έχει αποφασίσει το Σώμα των Επιτρόπων. Όμως, ο Επίτροπος έχει κάθε πρόθεση να το κάνει. Αυτή τη στιγμή θα έχει ληφθεί απόφαση από το Σώμα των Επιτρόπων. Καταλαβαίνουμε όλες αυτές τις επιθέσεις ε, κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις ε, συζητήσεις ε, με τους Αμερικανούς για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη για το θέμα αυτό. Επί του θέματος αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε τοποθετηθεί. Γνωρίζετε όμως ότι είχε τοποθετηθεί πολύ κατηγορηματικά σε σχέση με τους ε, γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τις ορμόνες. Ο πρόεδρος Παρόζο είχε πει ότι δεν θα είναι τμήμα των συζητήσεων ε, για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τι ΗΠΑ. Δεν θα συζητήσουμε για τι ορμόνες και τους γενετικώ τροποποιημένους οργανισμούς. Για την κλωνοποίηση δεν είχαμε συζητήσει ακόμη τότε, δεν είχε συζητήσει ακόμη τότε το Σώμα των Επιτρόπων. Δεν ήταν τμήμα τη συζήτηση με του ε, Αμερικανού. Αλλά δεν αποτελεί μυστήριο για κανέναν ότι οι Αμερικανοί πίεσαν πάρα πολύ όλα τα κρατη και εσάς ε, σίγουρα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφευχθούν ε, προτάσεις σε σχέση με την ετικετοθεσία ε, της πρώτης γενεάς κλώνων. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι προτάσεις που θα γίνουν θα βασιστούν σε επιστημονικά στοιχεία και στην ευημερία των ζώων. είναι σαφές ε, ότι η κλωνοποίηση έχει ως αποτέλεσμα θνησιμότητα, ε, δυσλειτουργία της ε, αναπαραγωγής, δημιουργεί και προβλήματα ευημερία των ζώων, είτε στις μητέρες είτε στους όσους συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία κλωνοποίησης. Ε, βάσει λοιπόν της ευημερία των ζώων θα υποβάλουμε και τις προτάσεις μας. Ε, βέβαια οι λόγοι αυτοί δεν υπήρχαν για την πρώτη γενεά, γιατί η πρώτη γενεά προκύπτει τουλάχιστον από τεχνητή γονιμοποίηση και δεν υπάρχει αυτό το θέμα της ευημερία των ζώων ε, για τα ζώα που προκύπτουν από την πρώτη γενεά. Οπότε θα ήθελα να ολοκληρώσω σε σχέση με αυτό που είπατε, δηλαδή ότι η συζήτηση θα είναι πολύ δύσκολη στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της ε, του Επιτρόπου Μπόρτζ ενώπιον του Κοινοβουλίου και τις οποίες επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Παρόσο στη συνέχεια. Όμως ε, η πρόταση ενδεχομένως ε, να μην σας βρει σύμφωνος ε, παρόλα αυτά. Ελπίζω να ε, χρήζει συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρχε κάποια στιγμή μια εναλλακτική επιλογή που είχε υπάρξει στον αέρα, ότι οι προτάσεις θα υποβληθούν για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Αποφασίστηκε από το Σώμα των Επιτρόπων να ε, υποβληθούν τώρα οι προτάσεις χαριντήρησης αυτών των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, χάρη σεβασμού βέβαια των ε, βουλευτών ε, που τόσο πολύ είχαν εμπλακεί σε αυτόν τον τριμερή διάλογο του 2011. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει παρόλα αυτά υπόψη τις ανάγκες ή τις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, επαναλαμβάνω, μπορεί να απογοητευτείτε από την έλλειψη φιλοδοξίας της πρότασης αυτής, η τις επιθυμιες του ευρωπαικου κοινοβουλιου όμως ήταν αντικείμενο πολύ δύσκολο συμβιβασμό στο πλαίσιο του Σώματος των Επιτρόπων. Πολύ δύσκολο συμβιβασμό. Και βεβαίως θα ε, εναπόκειται μετά στο συνομοθέτε, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, του Συμβουλίου και του Μελλοντικού Κοινοβουλίου και του Τωρινού Κοινοβουλίου, να ε, μπορέσουν να βρουν, να μπορέσουν να συμφωνήσουν επί του κειμένου αυτού. Βέβαια, αν πάλι αποτύχουν οι συζητήσεις αυτές, θα παραμείνουμε στην τρέχουσα κατάσταση που δεν απαγορεύεται το κλωνοποίηση. Δεν απαγορεύεται αυτή τη στιγμή η κλωνοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε πρόκειται για ερευνητικού λόγους, ε, για ενίσχυση των ε, ειδών προς εξαφάνιση κλπ είτε για ε, κρέας που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Δεν απαγορεύεται το η κλωνοποίηση, οπότε νέα αποτυχία των συζητήσεων θα διατηρήσει αυτή την κατάσταση, ε, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι ευνοϊκό για την ευημερία των ζώων. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έγινε η συζήτηση αυτή, παρά το γεγονός ότι βέβαια αισθάνθηκε ότι τις επιτέθηκαν πάρα πολύ, ε, επιτέθηκε πάρα πολύ η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω μια ακόμα ερώτηση να σας απευθύνω. Είπατε ότι είναι δύσκολο η Κομισιόν να απαντήσει σε μια επιστολή του Πρόεδρου μας, δεδομένου ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων ακόμα δεν έχει λάβει οριστική απόφαση. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείεται να ξεκινήσετε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για αυτό το θέμα πριν να γίνει η πολιτική συζήτηση μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν να ολοκληρωθεί η πολιτική συζήτηση. Λέτε ότι η Κομισιόν θα λάβει υπόψη την επιστημονική βάση που υπάρχει και θα τη θέσει ως βάση για τις διαπραγματεύσεις. Δεν πιστεύετε ότι ε, θα έπρεπε να εφαρμόσετε τα ίδια κριτήρια, δεδομένου ότι η συζήτηση είναι τόσο πολιτική που η Κομισιόν δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με τις ΗΠΑ για οποιασδήποτε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μέχρι ότου επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων για το θέμα της κλωνοποίησης των ζώων. Είναι δύσκολο να απαντήσω εγώ προσωπικά σε αυτήν την ερώτηση, Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι η εκκίνηση των διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ έγινε πριν από μερικούς μήνες. Η κλωνοποίηση τότε δεν ήταν τμήμα της συζήτησης. Αντίθετα με τις ορμόνες και τη, τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς για πράγματα, θέματα για τα οποία ο κ. Μπαρός έχει θέσει μια κόκκινη γραμμή στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Η κλωνοποίηση όμως τότε δεν αποτελούσε τμήμα της συζήτησης. Γιατί, Γιατί δεν είχε γίνει πολιτική συζήτηση για αυτό το θέμα στο Κολέγιο των Επιτρόπων και ε, ούτε και στο Συμβούλιο ή στο Κοινοβούλιο. Η αξία της πρότασης που θα είναι διαθέσιμη σε μερικές μέρες θα είναι ότι θα ξεκινήσει αυτήν ακριβώς τη συζήτηση ανεξάρτητα αν μας αρέσει η πρόταση ή όχι. Αντίθετα με το τι θα είχε συμβεί αν η Κομισιόν αποφάσιζε να αναβάλει τη συζήτηση και την υποβολή της πρότασης μέχρι το τέλος του 2014 για να γίνει αυτό ενόψη, ε, υπόψη του καινούργου κοινοβουλίου. Η Κομισιόν αποφάσισε να υποβάλει την πρόταση της τώρα προκειμένου να ξεκινήσει ακριβώς αυτή η συζήτηση και για την κλωνοποίηση αλλά και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, Συναρτήσει λοιπόν των ε, συζητήσεων που θα γίνουν για αυτήν ακριβώς την πρόταση που θα υποβληθεί σε μερικές μέρες δηλαδή αν την υιοθετήσει το Κολέγιο των Επιτρόπων την Τετάρτη, θα αποσταλεί Δευτέρα περίπου στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως να τη συζητάτε, να εκφράσετε την πολιτική σας θέση, όχι μόνο σε σχέση με το ίδιο το κείμενο, όσο και σε, αλλά όσο και, σε σχέση με τις ε, διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για αυτή την απάντηση. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Τροπολογίες μέχρι τις 8 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε θα έχει δημοσιευθεί και η πρόταση της Κομισιόν ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΜΒΙ στις 30 Ιανουαρίου του 2014 ενώ το ψήφισμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί σε μία ψελομέλεια του Φεβρουαρίου. Αυτά είναι τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Αύριο στις 9 ξεκινάμε με τη συνεδρία των συντονιστών και στις 10 ε, θα ξεκινήσουμε με την ε, υπόλοιπη ημερήσια διάταξη.